So, ladies uh, and uh, Κυρίες και κύριοι, καθυστερήσαμε δύο ακόμα λεπτά από την κανονική καθυστέρηση γιατί μετά από το μεσημεριανό διάλειμμα από ό,τι βλέπω δεν έχουν φτάσει και τόσα πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή την αίθουσα. Ωστόσο, καλωσορίζω τις δύο ομάδες των επισκεπτών στην Επιτροπή μας. Πρώτον, καλωσορίζω την αντιπροσωπεία από την Ιορδανία, τα μέλη του Ιορδανικού Κοινοβουλίου με επικεφαλής τον κύριο Σουλεϊμάν Αλσάμπατ Αντιπρόεδρο. Καλωσορίσατε στην Επιτροπή μας και καλή συνέχεια σας εύχομαι στην παραμονή σας εδώ. Και δεύτερον, Έχουμε κοντά μας μια ομάδα νέων ανθρώπων από τη Βόνη που ε, προσδοκούν να εργαστούν εδώ. Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας. So, one minute, ε, ένα λεπτό ακόμα θα περιμένουμε και δέκα θα ξεκινήσουμε. Good. Ωραία. Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινούμε τώρα την ε, απογευματινή μας συνεδρίαση επίσημα. Το πρώτο θέμα της ημερήσια διάταξη είναι το θέμα υπαριθών 15 και θα μιλήσουμε με τη Λετωνική Προεδρία για το τελευταίο εξάμεινο, τις επιτυχίες, και τα επιτεύγματα που είχαμε στον τομέα της ε, διεθνούς εμπορίου. Έχουμε μαζί μας την Κοινοβουλευτική Υπουργό για τις υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Λετωνίας. Σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά. Το τελευταίο εξάμεινο συζητήσαμε πολλά θέματα. Να σας υπενθυμίσω απλώς ενδεικτικά τα ζητήματα που σχετίζονταν με τους κανόνες για τις εισαγωγές, της χρηματοδοτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, την πρόοδο όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται εξέλιξη σε σχέση με διάφορες εμπορικές συμφωνίες, με το TTIP, με την Ιαπωνία, ε, με τα ε, περιβαλλοντικά προϊόντα Είχαμε ζητήματα που σχετίζονταν με τους μηχανισμούς και τα εργαλεία προστασίας του εμπορίου και την εμπορία προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και, για, ε, και στο πλαίσιο της ε, θανατικής καταδίκης. Είχαμε και κάποιες προόδους στο θέμα του TIP, δημοσιεύτηκε και εντολή αυτό που μας στενοχωρεί λίγο είναι το γεγονός ότι δεν υπεγράφει τελικά η σύμβαση για την διαφάνεια όσον αφορά τις ε, σχέσεις επενδυτών και κρατών. Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας στον τομέα αυτό με το Συμβούλιο. Υπάρχει λοιπόν μια ολόκληρη παλέτα θεμάτων με τα οποία ασχοληθήκατε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι εδώ στην Επιτροπή Ίντα για να συζητήσουμε ζητήματα που σχετίζονται με το εμπόριο. Για εμάς αυτά τα, αυτοί οι έξι μήνες της πρώτης Λετωνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν μια εξαιρετική και πολύ χρήσιμη εμπειρία. Από τον Ιανουάριο, όταν βρέθηκα εδώ για να σας παρουσιάσω τους στόχους της Λετωνικής Προεδρίας, επικεντρωθήκαμε στεναρά στο να καταστήσουμε την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική, πιο ψηφιακή και για να ενισχύσουμε τη συμμετοχή της στο διεθνή τομέα, προκειμένου να ε, επιφέρουμε θετικές αλλαγές για τους Ευρωπαίους πολίτες. Και χαίρομαι που είμαι στη θέση να σας πω ότι είχαμε πολλά επιτεύγματα καταλήξαμε σε συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων αλλά και για θέματα όπως είναι ε, το ξέπλυμα χρήματος και η εγγύηση για την νεολαία. Επίσης συνεχίστηκαν οι συζητήσεις για την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών, συζητοδρόμων και μέσω της στενής μας συνεργασίας με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τονίσαμε ότι η ανταγωνιστική Ευρώπη θα πρέπει να οικοδομείται στη βάση φιλόδοξων εμπορικών συμφωνιών και ότι θα πρέπει οι αποφάσεις μας να είναι διαφανείς προς τους πολίτες. Κατά τη διάρκεια της Λετωνικής Προεδρίας καταφέραμε να ε, έχουμε προόδους ε, όσον αφορά τις εμπορικές μας συμφωνίες με τρίτες χώρες. Και για πρώτη φορά στην ιστορία της Ένωσης επιδείξαμε υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας. Και καθώς οδεύουμε προς το τέλος της Λιτωνικής Προεδρίας θα ήθελα να σας περιγράψω ε, τι έχουμε επιτύχει στις εξωτερικές εμπορικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας ευχαριστήσω βεβαίως και για, την, ε, για το επικοδομητικό έργο των μελών της Επιτροπής Ίντα. Ήταν εξαιρετικά χρήσιμη η συμβολή σας στη διάρκεια των ε, φιλόδοξων διαπραγματεύσεων που είχαμε, αλλά και όσον αφορά το νομοθετικό έργο που έχουμε σε συνεργασία με το Συμβούλιο. Η οικονομική κρίση απέδειξε ότι το εμπόριο δεν ήταν ποτέ τόσο σημαντικό για την οικονομία της Ευρώπης όσο σήμερα. Ο νέος, η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εμπόριο συζητήθηκε για πρώτη φορά σε υπουργικό επίπεδο και στόχος μας είναι να αυξήσουμε την ανταγωνίστικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της σύναυσης νέων εμπορικών συμφωνιών προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε τις οικονομικές δυνατότητες και για να οριστικοποιήσουμε τις εμπορικές αυτές συμφωνίες. Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε ότι οι επενδύσεις και το εμπόριο αποτελούν εξαιρετικά χρήσιμα εργαλεία για την ανάπτυξη και την ε, αύξηση της απασχόλησης στην Ευρώπη. Περίπου 30 εκατομμύρια θέσεις εργασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω από το 14% της απασχόλησης, εξαρτώνται από το εμπόριο της Ένωσης με τρίτες χώρες. Αυτό ο αριθμός έχει πολλαπλασιαστεί σε σύγκριση με, τα προηγούμενα, με ό,τι συνέβαινε πριν από 20 ε, χρόνια. Επιπλέον ένα δισεκατομμύριο εξαγωγές σχετίζονται με τη διατήρηση 14.000 θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να περάσω τώρα στα ε, ζητήματα που σχετίζονται με το πολυμερές εμπόριο και το περιβάλλον. Η Προεδρία υποστήριξε πλήρως ένα διεθνές εμπορικό σύστημα προσπαθώντας να κατακτήσει ακόμη περισσότερη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με όλες τις πλευρές και τους εταίρους μας στον κόσμο. Προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε την ε, ε, κατάσταση μέσω της ε, ενίσχυσης και της εφαρμογής της συμφωνίας της Ντόχα και συγκροτώντας ένα πρόγραμμα εργασίας για την περίοδο μετά τον Παλί. Στη διάρκεια της Προεδρίας μας καλέσαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνενέσει στην Συμφωνία για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου. Οι κύριοι στόχοι της συμφωνίας είναι να απλωστευτούν οι τελωνιακές διαδικασίες και να εξασφαλιστεί ότι οι εμπορικές ροές είναι όσο πιο προβλέψιμες και ότι ολοκληρώνονται χωρίς προβλήματα. Σύμφωνα με τους δείκτες για τη διευκόλυνση του εμπορίου του ΟΣΑ, οι δείκτες αυτοί μάλλον εμπεριέχονται στη συμφωνία και μπορούν να αυξήσουν το ε, εμπόριο σημαντικά τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις αναπτυγμένες χώρες. Ελπίζουμε ότι οι εσωτερικές διαδικασίες για την κύρωση αυτής της συμφωνίας θα ολοκληρωθούν πριν από την υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ που θα γίνει στο Ναϊρόμπι. Πρόκειται για μια σημαντική απόφαση που θα συμβάλλει στην συνοριακή διακίνηση αγαθών, αλλά θα αποτελέσει και μια σημαντική βάση για τη διαπραγματεύση στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Ντόχα. Το άτυπο Συμβούλιο Εμπορίου στη Ρήγα συνέβαλε στον επικοδομητικό διάλογο για την κατάσταση και τη διαδικασία μετά το Μπαλί. Οι Υπουργοί Εμπορίου εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην Τόχα και επίσης εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς, τον, προς τις προσπάθειες του ΠΟΕ προκειμένου να επιτευχθεί σύγκληση μεταξύ των μελών του ΠΟΕ προκειμένου να ολοκληρωθεί η αναπτυξιακή αντέντα της Ντόχα εν ώψη και της διάσκεψης στο Ναϊρόμπι. Στην ε, ε, συνάντηση αυτή που έγινε στις 7 Μαΐου εκφράστηκε και στεναρή υποστήριξη για το πρόγραμμα εργασιών μετά το Μπαλί και επιβεβαίωσε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να βρεθεί μια ρεαλιστική προσέγγιση για το μέλλον. Μια άλλη διαδικασία που σχετίζεται με την ε, ενίσχυση της ε, πολυμερού, του πολυμερού συστήματος εμπορίου αφορά τις προσχωρήσεις σε εμπορικές συμφωνίες και είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι οριστικοποιήθηκαν οι διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση του, Καζαστάν, του Καζακστάν και κρεμεί μόνο η επίσημη κύρωση του, της ε, συμφωνίας. Επίσης, υποστηρίξαμε την σύναψη συμφωνίας για τις ε, υπηρεσίες, για τα περιβαλλοντικά προϊόντα, καθώς και συμφωνία ε, για τα προϊόντα πληροφορικής. Όσον αφορά την ε, διμερή ατζέντα εμπορίου, θα ήθελα να τονίσω την ε, σημασία που έχουν οι διμερείς εμπορικές συμφωνίες, με παράδειγμα την Νότιο Κορέα. Τα τρία χρόνια αυτά που η συμφωνία βρίσκεται σε ισχύ, οι εξαγωγές οχημάτων προς την Νότια Κορέα έχουν αυξηθεί κατά 90%, ενώ οι νοτιοκορεατικές επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν από 13 δις το 10 σε 18 δις το 2012. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ σε μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες όσον αφορά τις επενδύσεις ε, και το εμπόριο στη διάρκεια της Λετωνικής Προεδρίας την Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων. Και χαιρόμαστε που στη διάρκεια της Προεδρίας μας υπήρξε κινητικότητα όχι μόνο όσον αφορά τη διαφάνεια, αλλά και τη συμμετοχή στη συζήτηση των ενδιαφερόμενων μερών και τη κοινή γνώμη. Είμαστε ικανοποιημένοι που υπήρξε σταθερή πρόοδος στη διάρκεια των δύο τελευταίων ε, κύκλων διαπραγμάτευσης και επίσης είναι σημαντικό να συνεχιστεί το έργο για τη διευκόλυνση των ευκαιριών που προσφέρονται σε μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, στη Λετωνία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιστοιχούν στο, σε πάνω από το 50% των εξαγωγών προς τη ΣΥΠΑ. Παρόλα αυτά όμως, πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν ακόμη εμπόδια όσον αφορά τις εξαγωγές τους προς τη ΣΥΠΑ, τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της συμφωνίας TTIP. η επιτυχής ε, ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το TTIP μπορεί να ε, υπάρξει μόνο σε περίπτωση που τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργαστούν επιτυχώς. Δεν θα πρέπει να στέλνουμε μεικτά μηνύματα στους ομολόγους μας για το τι θέλει να πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις διαπραγματεύσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι μια κατάλληλη λύση μπορεί να βρεθεί για θέματα τα οποία προκάλεσαν ευρεία συζήτηση. Η Λετωνική Προεδρία παραμένει πεπισμένη ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία για, μια, ε, για ένα μεταρρυθμισμένο μηχανισμό επίλυσης διαφορών κρατών και επενδυτών στο TTIP. Έγινε σημαντική δουλειά επί της Προεδρίας μας για να μεταρρυθμίσουμε τον μηχανισμό προστασίας των επενδυτών. Το Συμβούλιο ε, εξέτασε το έγγραφο ISDN ε, που παρουσιάστηκε το Μάιο από την Κομισιόν στην Επιτροπή, την Αρμόδια, ως βάση για να υπάρξει μεταρρύθμιση αποδεκτή από όλους τους εμπλεκόμενους. Στους επενδυτικούς κανόνες ε, δεν θα πρέπει να υπάρχει περιορισμός των δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών να ρυθμίζουν θέματα δημοσίου όπως είναι υγεία, ασφάλεια, ε, προστασία των καταναλωτών, περιβάλλον, προστασία των δεδομένων και κάποια άλλα. Υπάρχει σαφής ε, σύγκληση απόψεων ότι το δικαίωμα ε, ρύθμισης θα πρέπει να απεικονιστεί ε, μέσω μέτρων δηλαδή, θα πρέπει να απεικονιστεί στην συμφωνία. Ω Προεδρία έχουμε ισχυριστεί πάντα ότι μια επιτυχής ολοκλήρωση τη της εταιρικής σχέσης με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού θα έχει οικονομικά ωφέλη και θα προωθήσει τις κοινέ μας αξίες. Ενώ υπάρχουν μεγάλες βελτιώσεις ε, στην επικοινωνία μα με το κοινό, πιστεύουμε ότι οι και μερικές φορές ε, κάποια εχθρότητα που υπάρχει στην κοινή γνώμη θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με πληροφόρηση και με ανοιχτό διάλογο. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να παίξουν εδώ κάποιο ρόλο. Αγαπητοί βουλευτές, επιτρέψτε μου τώρα με δύο λόγια να μιλήσω για άλλα σημαντικά θέματα που αφορούν τις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Όπως ξέρετε, μια σημαντική πρόοδος έχει επιτεθεί στις διαπραγματεύσεις εμπορικές με το Βιετνάμ και την Ιαπωνία. Η Κορυφή τη Ευρωπαϊκή Ιαπωνίας τέλος του Μαΐου στο Τόκιο ήταν ε, η κατάλληλη όθηση για να διευκολυνθούν οι διαπραγματεύσεις και να επιταχυνθούν οι, προσπάθειε μα μας για να πετύχουμε μια ε, φιλόδοξη συμφωνία κυρίως για μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά και για τις δημόσιε συμβάσεις. Οι διαπραγματεύσεις ε, ελευθερών εμπορίου με το Βιετνάμ μπήκαν σε μια εντατική τελική φάση με τις διαπραγματεύσεις πολύ πιθανόν να ολοκληρωθούν στο εγγύ μέλλον. Είναι σημαντικό να αναπτύξουμε περαιτέρω τις εμπορικές σχέσεις με την Νοτιοανατολική Ασία. Όπω αναγνώρισε και η επίτροπο Μάλστρομ στην Σύνοδο Κορυφή ΑΣΕΑΝ, το, υπάρχει το δυναμικό για να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία ε, και σε πολυμερή και σε διμερή βάση. Η επερχόμενη σύνοδος κορυφής με την Κίνα θα αποτελέσει μια ευκαιρία να αν, ξαναδούμε τις διαπραγματεύσεις για μια συνολική συμφωνία για τις ε, επενδύσεις με την Κίνα, ε, να εκφράσουμε τις φιλοδοξίες μας για την διαφάνεια, ε, ένα αξιόπιστο καονιστικό πλαίσιο, βιώσιμη ανάπτυξη και πρόσβαση αγορά. για να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει που αντιμετωπίζουν οι εταιρείε μα στην κινέζικη αγορά. Το πρώτο σημαντικό βήμα στι σχέσει μα θα πρέπει να είναι η ολοκλήρωση της επενδυτική συμφωνία. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν να ολοκληρώσω θα ήθελα σύντομα να στραφώ σε μία από τι σημαντικέ προτεραιότητε τη Λεδονικής Προεδρία, την ενίσχυση των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων με τους ανατολικού μας γείτονες και εταίρους. Η Λετωνική Προεδρία, σε στενή συνεργασία με την Κομισιόν, διοργάνωσε την πρώτη υπουργική συνάντηση για το εμπόριο ε, με τα μέλη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Ε, οι Υπουργοί Εμπορίου συναντήθηκαν με τους ομολόγους από την Αρμενία, Αζερβαϊτζάν, ε, Λευκορωσία, Γεωργία, Μολδαβία και Ουκρανία και μελέτησαν τις δυνατότητε που υπάρχουν για την ανάπτυξη ε, μια εμπορική διάσταση στην εταιρική σχέση. Η προσωρινή εφαρμογή του DCFTA δίνει αποτελέσματα. Στην περίπτωση τη Μολδαβία βλέπουμε ότι το 2014 οι εξαγωγέ στη Μολδαβία αυξήθηκαν κατά 3%, ενώ οι εισαγωγέ από τη Μολδαβία αυξήθηκαν κατά 20%. Το DCFTA, η εφαρμογή αυτή τη συμφωνία δηλαδή, ε, περιλαμβάνει ένα πλήρες πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, ούτως ώστε να φέρει πιο κοντά τις χώρες Μολδαβία και Γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό αυτή η μεταρρύθμιση να συνεχιστεί σε αυτές τις χώρες και να έχουν οι χώρες αυτές ε, απτά ωφέλη από το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίγουσες μεταρρυθμίσεις απαιτούνται στην Ουκρανία επίσης. Το μνημόνιο συνεννόησης ε, που μιλάει για το πρόγραμμα πολιτικής προσαρτισμένο στο νέο μακροοικονομικό πρόγραμμα βοήθειας, θα υποστηρίξει την μεταρρυθμιστική ατζέντα που προωθούν οι Ουκρανικές αρχές για πολλούς τομείς. Οι σύνος κορυφή τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ουκρανία επιβεβαίωσαν ότι η προσωρινή εφαρμογή τη συμφωνία με την Ουκρανία DCFTA θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2016. Και η υπουργική συνάντηση με τους ανατολικούς εταίρους για το εμπόριο και η σύνος με τους ανατολικούς γείτονες μίλησαν για την, ε, τόνισαν την σημασία περαιτέρω ανάπτυξη μιας επιτυχούς εμπορικής διάστασης στην ε, εταιρική σχέση με, τους, με τους, ε, τις χώρες αυτές ως πηγή ανάπτυξης θέσεων απασχόλησης σε αυτές τις χώρες. και εμείς δείξαμε ότι είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε για τέτοιες εμπορικές σχέσεις. Και τέλος, θα ήθελα σύντομα να αναφερθώ σε κάποιους νομοθετικούς φακέλους. Θα ήθελα να, να δώσω έμφαση στην καλή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδήγησε σε γρήγορη υιοθέτηση ε, φακέλων για μεταρρύθμιση <clears throat> για μέτρα εποπτείας και διασφάλισης για τις εισαγωγές κλώστο υφαντουργικών και άλλων προϊόντων από χώρες που δεν είναι μέλη του ΠΟΕ. Αυτές είναι δύο προτάσεις ε, που κληρονομήσαμε από το τρίο, ε, από τον εταίρο μας μάλλον στο τρίο, την Ιταλική Προεδρία και συνεχίσαμε εμείς και την προωθήσαμε. Ε, θέλουμε καταρχάς στην νομοθετική πρόταση αυτή να έχουμε ένα ενωσιακό σύστημα για την αυτοπιστοποίηση των υπεύθυνων εισαγωγέων μεταλλευμάτων από περιοχές πολέμου ε, το συζητήσαμε στο Συμβούλιο και στην ομάδα εμπειρογνωμόνων. Ε, ευχαριστούμε το Κοινοβούλιο για τη δουλειά Θα πρέπει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να συνεχίσουν την εξέταση του φακέλου. Κατά τη διάρκεια τη Προεδρία μα, είχαμε έντονε συζητήσει στο Συμβούλιο για τον κανονισμό που απαγορεύει το εμπόριο κάποιων αγαθών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια ή άλλε ε, απάνθρωπες, ε, και ε, συμπεριφορέ. Ε, μεταχείριση ή τιμωρίες. Θέλουμε να δούμε και την πρόταση του Κοινοβουλίου για αυτό το θέμα. Τελειώνει η Προεδρία μας, αλλά η δουλειά για αυτές τις εμπορικέ προτεραιότητες θα συνεχιστούν. Περιμένουμε να συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή τα κυρίω. για να συνεχίσουμε τη δουλειά που, έχουμε, που κάνουμε και να βελτιώσουμε την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρεμβαίνει σε παγκόσμια κλίμακα. Γι' αυτό η Προεδρία μας ε, θέλει να ε, ευχηθεί στους διαδόχους μας που είναι το Λουξεμβούργο. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε Υπουργέ που μας κάνετε αυτή την πλήρη και εξαντλητική παρουσίαση της, ε, των εργασιών σας. Θα δώσω τώρα το λόγο στις πολιτικές ομάδες. Ο Ντανιέλ Κασπάρη από το ΕΛΚ πρώτος. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Δύο σύντομες ερωτήσεις θα ήθελα να θέσω. Νομίζω ότι σκιαγραφίσατε πολλά ζητήματα και αναφερθήκατε σε αρκετές επιτυχίες. Θέλω όμως να σταθώ σε δύο σημεία. Πρώτον, αναφερθήκατε στην ανατολική γειτονία και στο θέμα της Ουκρανίας. Πιστεύετε ότι η κατάσταση στο Συμβούλιο θα παραμείνει τόσο σταθερή όσο στο Κοινοβούλιο, ότι θα επιμείνει δηλαδή να τεθεί σε ισχύ ε, το αργότερο πρώτης πρώτου του 16 100% χωρίς νέες υποχωρήσεις αυτή η συμφωνία για, την, ε, για το ελεύθερο εμπόριο ή θα υπάρξει πρόβλημα. Και δεύτερον, δεν αναφέρατε δύο πράγματα. Την το εργαλείο IPI και τη μεταρρύθμιση TTIP. για την πρόσβαση στην αγορά. Είναι θέματα που θα παραδώσετε στην επόμενη Προεδρία ή χάθηκαν κάπου στο δρόμο. Έχετε κάποια ιδέα για το ποια θα είναι η θέση του Συμβουλίου για το φάκελο για ε, τα ε, ορυκτά που προέρχονται από ζώνες σύγκρουσης. Uh, Παρακαλώ. Τέσσερις παρατηρήσεις. Η πρώτη σχετίζεται και με το πρώτο ερώτημα του κυρίου Κασπάρη για την Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας, μας ενημέρωσε ότι στις 13 Ιουνίου η Ρωσική Ομοσπονδία παρουσίασε μια νέα πρόταση για τριμερή διάλογο. για το θέμα της Ουκρανίας. Ενδεχομένως υπάρχουν κάποια στοιχεία αντιφατικά και υπάρχει και αλληλοεπικάλυψη. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό. Δεύτερον, αναφερθήκατε στην Κίνα και τις επενδύσεις. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την πρόσβαση στην αγορά, με την αγορά, με την οικονομική κατάσταση της Κίνας. Άλλωστε, οι νομικές υπηρεσίες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεξεργάζονται το, το θέμα αυτό. Ποια είναι η γνώμη σας. Και τρίτον, δεν μιλήσατε για τις στατιστικές για το εξωτερικό εμπόριο. Για το φάκελο αυτό, ο οποίος ε, έφτασε σε ένα ικανοποιητικό σημείο στην Ιταλική Προεδρία και έκτοτε δεν έχει γίνει κάτι. Και τέταρτον να πω ναι υπάρχει περισσότερη διαφάνεια, έχει δημοσιευθεί και η εντολή για το TTIP και η εντολή για την TISA. Δεν θα έπρεπε αυτό να ισχύει για όλες τις εντολές που έχει το Συμβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Σάραλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κυρία Υπουργέ για την περιγραφή που κάνατε των καθηκόντων που δεν ήταν καθόλου εύκολα κατά τη διάρκεια της δικής σας προεδρίας. Πράγματι βρεθήκατε ενώπιον μιας περίπλοκης κατάστασης και καλώς ε, υπογραμμίσατε ότι ήταν αυτή μια περίοδος πάρα πολλών διαπραγματεύσεων και κυρίως διμερών εμπορικών συμφωνιών οι οποίες ήταν αντικείμενο επεξεργασίας. Γνωρίζουμε όλοι ότι παγκοσμίω και σε πολυμερές επίπεδο οι εξελίξεις έχουν κάπως παγώσει και έγινε αυτός ο αγώνας μεταξύ των χωρών για το ποια χώρα θα συνάψει και θα ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις πρώτη και γρηγορότερα από τις άλλες για διμερείς συμφωνίες και όχι πολυμερείς. Έτσι έχει κατάσταση, θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Και πράγματι συμφωνώ και εγώ ε, ότι η Προεδρία σας ήταν επιτυχημένη ως προς αυτό. Ε, καλωσορίζω τα σχόλιά σας για το TTIP, το οποίο δεν ήταν και το πιο εύκολο θέμα, ούτε καν στη δική μας Επιτροπή. Και περιμένουμε σύντομα να ξανασυζητηθεί το θέμα εδώ στην Επιτροπή μας. Ήθελα να κάνω μια παρατήρηση, η οποία είναι και ερώτηση συνάμα, γιατί αναφερθήκατε επανελειμμένως στα θέματα της διαφάνειας. Επομένως σας ερωτώ το εξής. Έχει σημειωθεί πρόοδος ή μπορούμε να περιμένουμε ότι θα σημειωθεί πρόοδος για το θέμα της εξέτασης ε, των συνθήκων. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Chair, and... Επόμενος ομιλητής, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ κυρία Υπουργέ για τις παρατηρήσεις σας. Προσπαθήσατε να προωθήσετε μεταρρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Είναι σαφές σε όλους μας ότι ε, δεν μπορεί μία μόνη Προεδρία να ε, ολοκληρώσει με μια μεταρρύθμιση είναι μια συνέχεια, είναι δουλειά συνέχειας και τα βασικά ζητήματα παραμένουν επιτάπητος. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, ποιο λιθαράκι είναι αυτό που μπορεί η Λετωνική Προεδρία να βάλει και που κατάφερε να βάλει. Αυτό εμένα με ενδιαφέρει να δω και έρχομαι λοιπόν στη σύμβαση ΣΥΤΑ. Μιλήσατε για το ISDS, για την παρουσίαση της νέας πρότασης από την Επίτροπο Μάλστρομ. Τι σημαίνουν όλα αυτά για τη Συμφωνία ΣΥΤΑ. Ξέρουμε ότι οι θέσεις των κρατών μελών είναι διαφορετικές ως προς την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας βάσει της έκβασης ε, των συζητήσεων του TTIP και της ρήτρα ISDS εκεί. Δεύτερον, η μεγαλύτερη από τις προκλήσεις είναι η σχέση μας με τις ε, χώρες που ανήκουν στην ανατολική γειτονία, στην πολιτική αυτή. Ο Πρόεδρος ήδη μας ενημέρωσε για την ε, ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόταση της Ρωσίας για την συνέχιση του τριμερούς διαλόγου, τον οποίο επιδιώκει η Ρωσία να επινοήσει. Ξέρω ότι τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές θέσεις. ως προς τον τρόπο με τον οποίο μελλοντικά θα διαμορφώσουμε τις σχέσεις μας με τη Ρωσική Ομοσπονδία ενώ από την άλλη θα εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας με τις χώρες που ανήκουν στην ε, πολιτική ανατολικής γειτονίας. Επομένως, οι εμπορικές συνομιλίες με τη Ρωσία πώς είναι δυνατόν να θεωρούνται πιθανές και να έχουμε λύσεις για το σύστημα των κυρώσεων που έχει επιβάλει Ε, ε. Πώς όλα αυτά ταιριάζουν μεταξύ τους και πώς μπορούν να μεταφραστούν σε συγκεκριμένα βήματα ούτως ώστε να πάυσει το οικονομικό και άλλο αδιέξοδο που έχουμε με τις ε, χώρες που ανήκουν στην Ανατολική ε, γειτονία. Αυτό ισχύει και για την Ουκρανία και για τη Μολδαβία και προσπαθούμε να υιοθετήσουμε και συγκεκριμένη θέση για την Γεωργία, το Αζερβαϊτζάν και την Αρμενία. Και δεν μιλήσατε και για τη σύνοδο ΣΕΛΑΚ με ε, τις χώρες της Λατινικής Αμερικής Καραϊβικής. Ποιες είναι οι δυνατότητες εμπορικής συνεργασίας και συνέχισης των εμπορικών διαπραγματεύσεων με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής για την ε, εμπάθηση της ολοκλήρωσής μας με αυτές τις χώρες. Ευχαριστώ. κυρία ευχαριστώ. Να προσθέσω και εγώ κάποιες, ε, κάποια πράγματα στις ερωτήσεις που τέθηκαν ήδη. Για το ΣΥΤΑ, θα ήθελα να μάθω αν από τη δική σας, ε, κατά τη γνώμη η απο πλευρα ήδη οριστικοποιηθεί ε, ή αν θα υπάρξουν μικρές αλλαγές. Για το ISDS ε, αναφερθήκατε στις συζητήσεις που υπήρξαν στο Συμβούλιο σε σχέση με την πρόταση Μάλστρομ. Υπήρξε όμω και η πρόταση του κυρίου Γκάμπριελ και θα ήθελα να μάθω τι συζητήθηκε επί της συγκεκριμένη πρόταση στο Συμβούλιο. Υπάρχει πλειοψηφία για το δικαστικό σύστημα που ε, πρότεινε εκείνος για τα, για τα που προέρχονται από ζώνε συγκρούσεων. Θα ήθελα να μου πείτε αν θα θέλατε να ξεκινήσει ο τριμερής διάλογος τώρα, επί δική σας ε, προεδρίας, ή αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό, και τέλος ε, θέλω και εγώ να τονίσω το ζήτημα της ε, διαφάνειας της ε, εντολής. Θεωρώ ότι το Συμβούλιο μπορεί να προχωρήσει και να δημοσιεύσει όλες τις εντολές που έχει όσον αφορά τις εμπροϊκές διαπραγματεύσεις τις οποίες προβαίνει. Υπάρχουν συζητήσεις για αυτό το θέμα, έχουν εκφραστεί αντιρρήσεις και ανέα ποιον. Ωραία, δεν έχει ζητήσει κάποιο άλλο το λόγο λέει ο Πρόεδρος. Επομένως, Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για τα ερωτήματα και για τα σχόλιά σας. Και για το γεγονός ότι εκφράσατε τις απόψεις σας και ότι εκφράσατε τις ε, ανησυχίες σας για πολλά από τα ζητήματα. Και χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να δώσω επαντήσεις και να σας περιγράψω τι έχουμε επιτύχει διεξοδικότερα. Όσον αφορά τις συζητήσεις ε, στο Συμβούλιο, Εργαζόμαστε σκληρά για να σημειωθεί πρόοδος. Όπως είπατε κι εσείς και όπως γνωρίζετε, τα θέματα συζητώνται από Προεδρία σε Προεδρία. Πάντως, στα ε, ζητήματα που είχαμε επιλέξει, προσπαθήσαμε να τα αποκρισταλώσουμε και σε, σε συγκεκριμένα οικονομικά πλεονεκτήματα. Τα περισσότερα ερωτήματα που τέθηκαν ε, αφορούσαν το τίτυπο, οπότε θα ξεκινήσω με αυτό το θέμα. Θα ήθελα, λοιπόν, να τονίσω ότι δεν πρόκειται απλά για μια εμπορική συμφωνία με πολλές δυνατότητες για την ανάπτυξη της οικονομίας. Αποτελεί και μια συμφωνία που θα ενισχύσει τη στρατηγική μας εταιρική σχέση με τις ΗΠΑ. Και αυτή ήταν πάντοτε η οπτική από την οποία εμείς ως Ελληνική Προεδρία ε, προχωρούσαμε στις διαπραγματεύσεις. Φυσικά και θέλουμε να έχουμε και οικονομικά ε, πλέον και για να γίνει κάτι τέτοιο η συμφωνία θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και φιλόδοξη. Και αντί να διαγράφουμε θέματα από την ε, ημερήσια διάταξη και ε, από τον κατάλογο των συζητήσεων θα έπρεπε να κάνουμε το αντίθετο. Για το ISDS, όπως είπα και νωρίτερα, θεωρούμε ότι το έγγραφο που παρουσίασε η Επίτροπος Μάλστρομ αποτελεί μια θετική βάση για την μεταρρύθμιση του συστήματος, αλλά έχουν εκφραστεί διάφορες ανησυχίες όσον αφορά το σύστημα ISDS. Και στο πλαίσιο αυτό ε, ρωτήσατε και για την ε, Συμφωνία ΣΥΤΑ. Πιστεύω ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι συζητούμε μια συμφωνία, τη Συμφωνία ΣΥΤΑ, που έχει ήδη συναυθεί. Άρα υπάρχουν δυνατότητες περιορισμένες ε, για να αντιμετωπιστούν ορισμένα νομοθετικά νομικά ζητήματα και θα πρέπει αυτό να γίνει σε συμφωνη... με, με τη σύμφωνη γνώμη και της καναδικής πλευράς. Από αυτή την άποψη λοιπόν ε, το ζήτημα της συγκεκριμένης συμφωνίας έχει κλείσει. Αλλά όσον αφορά την διαφάνεια, πιστεύω και εγώ ότι είναι πράγματι το πιο σημαντικό ζήτημα και ήταν το πιο σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίσαμε εμείς στη διάρκεια αυτών των έξι μηνών και είμαι περήφανη που σημειώθηκε σημαντικότατη πρόοδος στο θέμα της διαφάνειας. Οι διαπραγματευτικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δημοσιευθεί στο διαδίκτυο μαζί και με διάφορες άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες ε, συζητήσεις. Και πολλοί ευρωβουλευτές έχουν δηλώσει ότι έχουν πλέον πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που χρειάζονται και για τα οποία ενδιαφέρονται. Άρα η διαφάνεια είναι ένα σημαντικότατο στοιχείο για να προχωρήσουμε από εδώ και στο εξή. Και εμεί, ω Λετωνική Προεδρία πάντοτε θεωρούσαμε εξαιρετικά σημαντική τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, τη κοινωνία των πολιτών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην όλη διαδικασία. Η διαφάνεια λοιπόν είναι σημαντική και είναι σημαντικό ότι οι πολίτε και οι οργανώσει του έχουν πλέον περισσότερη πρόσβαση σε πληροφορίε προκειμένου και εμείς να είμαστε βέβαιοι ότι οι διαπραγματεύσεις ε, διεξάγονται ε, με διαφάνεια απέναντι σε, όλους, σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και θεωρώ ότι η διαφάνεια σε εμπορικές διαπραγματεύσεις θα πρέπει να αποτελέσει μια ε, σημαντικότατη αρχή γιατί η συμμετοχή των πολιτών, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των κοινωνικών εταίρων το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει είναι να ενισχύσει τη θέση μας προκειμένου να βρίσκουμε τις καλύτερες λύσεις και να συνάπτουμε τις καλύτερες δυνατές συμφωνίες με άλλες χώρες. Ελπίζω λοιπόν ότι στο μέλλον θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες, ακόμα πιο επιτυχή αποτελέσματα όσον αφορά τη διαφάνεια και νομίζω ότι το TTIP αποτέλεσε μια καλή αφετηρία όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Για τα άλλα ερωτήματα που τέθηκαν, για τη συμφωνία με την Ουκρανία και την ανατολική εταιρική σχέση. Όταν μιλούμε για την Ουκρανία, δεν έχουμε κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι η θέση του Συμβουλίου θα αλλάξει. Το Συμβουλίο ε, πιστεύει ότι το TCFCA θα εφαρμοστεί από 1η Ιανουαρίου του 2016. Και στη διάρκεια της διάρκειας της Ρήγα εκφράστηκε στεναρή υποστήριξη και απόλυτη βεβαιότητα ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί την 1η Ιανουαρίου 2016. Βεβαίως έχουμε σημειώσει την πρόσφατη ρωσική πρόταση και ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει κανείς να λαμβάνει υπόψη του είναι ότι πρόκειται για διαπραγματεύσεις με αναξάρτητο κράτος, την ε, Ουκρανία. Μπορούν δηλαδή να συμμετέχουν στη συζήτηση, αλλά δεν έχουν δικαίωμα βέτο, άσκησης βέτο στις διαπραγματεύσεις. Άρα οι τριμερείς ε, συζητήσεις για την DCFDA θεωρούμε ότι, σε, ότι η πρόταση της ε, Επιτρόπου Μάλστρομ ήταν εξαιρετική βάση και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι κανείς δεν μπορεί να θέσει εμπόδια στη διαδικασία αυτή. Επίσης, ρωτήσατε για τις εμπορικές μας σχέσεις με τις ε, χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες να υπάρξουν στενότερες εμπορικές σχέσεις και με τη Μολδαβία και με τη Γεωργία και με τις υπόλοιπες χώρες και πιστεύουμε επίσης ότι μπορούμε να ε, βοηθήσουμε και ο ένας τον άλλον ε, και στο θέμα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και στα προβλήματα που έχουν προκύψει. Ο δρόμος που θα ακολουθήσουμε είναι η εφαρμογή των συμφωνιών που έχουν ήδη συναυθεί και η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που έχουν προκύψει από τις ενισχυμένες εμπορικές μας σχέσεις με αυτές τις χώρες. Για την Ασία τώρα και συγκεκριμένα να σας πω για την Κίνα. Το ερώτημα που έθεσε ο κύριος Λάγκε. Συμφωνώ απόλυτα ότι χρειάζεται να γίνουν περισσότερα πράγματα για να ενισχυθεί η συνεργασία μας με την Κίνα που πλέον αποτελεί και αναπόσπαστο στοιχείο των ε, στρατηγικών ανάπτυξης πολλών ε, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Στόχος μας είναι να διευρυνθούν οι εμπορικές ε, σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη συγκεκριμένη χώρα και παρά το γεγονός ότι το οικονομικό μοντέλο της Κίνας πράγματι θέτει ορισμένα προβλήματα δική μας επιδίωξη είναι να έχουμε μακροπρόθεσμες υγιείς σχέσεις με τη συγκεκριμένη χώρα. Όσον αφορά την κατάσταση, όσον αφορά την οικονομία της αγοράς στην Κίνα, μπορεί η συζήτηση να ξεκινήσει στη βάση, στο Συμβούλιο, στη βάση της πρότασης της Κομισιόν και θα πρέπει να υπάρξει σαφής αντίληψη για το ποιες θα είναι ε, οι, εμπορικές, ε, ε, οι νομικές επιπτώσεις της προσχώρησης της Κίνας στην, ε, ε, στον ε, Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Όσον αφορά την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πληροφορίες για τις διαπραγματεύσεις, για τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, το Συμβούλιο θα εξακολουθήσει να εξετάζει το θέμα αυτό κατά περίπτωση. Και κάθε αίτημα που υποβάλλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να αποκτά πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που σχετίζονται με τις διαπραγματεύσεις θα εξετάζεται στη βάση της κείμενης νομοθεσίας. Αλλά η γενική αρχή που ανέφερα και νωρίτερα είναι ε, αυτή της ε, γενικής διαφάνειας. Τώρα, για τα ορυκτά που προέρχονται από προ... ζώνες συγκρούσεων. Το Συμβούλιο κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες ε, για το συγκεκριμένο ζήτημα στη διάρκεια της Λετωνικής Προεδρίας και το θέμα αυτό συζητήθηκε και στο Συμβούλιο και μάλιστα υιοθετήθηκε και η προσέγγιση που πρότεινε η Κομισιόν. Στη διάρκεια της Προεδρίας μας ε, καταλήξαμε και συμφωνήσαμε στην γενική προσέγγιση για το ζήτημα αυτό για τα ε, ανακυκλώσιμα ε, προϊόντα, για τα προϊόντα εξόρυξης, για τα μεταβατικά μέτρα και για την, ε, τον, την, την, τη μεταχείριση του χρυσού ως ε, ορυκτού όταν δεν έχει περάσει από διαδικασία κατεργασίας. Τέθηκε κι άλλο ένα ερώτημα. Η Κομισιόν σημείωσε στο πρόγραμμα εργασιών της ότι η πρότασή της θα τροποποιηθεί φέτος προκειμένου να απλουστευτεί η διαδικασία, προκειμένου να μειωθούν οι ε, προθεσμίες για τις ε, ε, έρευνες. Όταν λοιπόν λάβουμε τις τροποποιήσεις θα ολοκληρωθούν και οι συζητήσεις στο Συμβούλιο. Τώρα για τα εργαλεία τα αμυντικά εργαλεία για το εμπόριο θα συνεχιστεί η εξέταση του θέματος και ελπίζουμε ότι η Κομισιόν θα ε, υποβάλει προτάσεις που θα αμβλύνουν τις, ε, τη διάσταση απόψεων που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών και δεν είναι μυστικό ότι τέτοια διάσταση υπόψεων υπάρξει. Και τέλος, να αναφερθώ και στη σύμβαση του ΟΗΕ για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο. Συζητήσαμε εκτενώς για το, το θέμα αυτό στην, στο Συμβούλιο ε, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ενεργειακά ζητήματα, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερο χρήματα. Η σύμβαση αυτή ε, είναι ανοιχτή προς κύρωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσχωρήσει οποιαδήποτε στιγμή θέλει και νομίζουμε ότι είναι σωστό και σόφρον να καταλήξουμε σε κοινή θέση και γι' αυτόν τον λόγο η Λετωνία δεν ε, εξέτασε ούτε προώθησε την, ε, την ε, προσχώρησή της ε, σε μεμονωμένη βάση στη συγκεκριμένη σύμβαση. Σταματώ εδώ. Για τη Λατινική Αμερική υπήρξε συνάντηση του Συμβουλίου, συζητήθηκε το συγκεκριμένο ζήτημα, το εμπόριο δηλαδή με οι εμπορικές σχέσεις με τη Λατινική Αμερική και είμαστε βέβαιοι ότι θα σημειωθεί πρόοδος και όπως ανέφερα και στην αρχή της τοποθέτησής μου, το εμπόριο είναι ένας από τους ε, πιο σημαντικούς ε, μηχανισμούς που έχουμε για να βοηθήσουμε την ανάπτυξη χωρών και για να κατακτήσουμε, να επιτύχουμε πλεονεκτήματα για τις πολίτες της Ένωσης. Οπότε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής ΙΝΤΑ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνδρομή σας στη διάρκεια αυτών των έξι μηνών της Λετωνικής Προεδρίας. Τα επιτεύγματά μας θα ήταν αδύνατα αν δεν είχαμε την ε, αποτελεσματική συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είμαι βέβαιη ότι θα συνεχιστεί αυτή η στενή συνεργασία και ότι το Συμβούλιο θα, θα συνεχίσει να ε, συζητά και να εξετάζει όλα αυτά τα ζητήματα που είναι ανοιχτά αλλά και τα μελλοντικά. Και ε, πιστεύω ότι το Συμβούλιο θα είναι πάντοτε πρόθυμο να βρίσκεται σε στενή συνεργασία και επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ήταν πολύ καλή συνεργασία. Πάντα ήσασταν στη διάθεσή μας. Είχατε ευήκο Προσπαθήσατε να βρείτε καλές λύσεις. Η συνεργασία ήταν άψογη. Καλή τύχη λοιπόν στη συνέχεια και προσωπικά και επαγγελματικά και προσωπικά. Και θα είμαστε πάντα σε επικοινωνία βέβαια. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα περάσουμε τώρα στο θέμα 16. Η πρώτη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον προπολογισμό της επόμενης χρονιάς. Γνωρίζετε ότι η Κομισιόν στις 27 Μαΐου υπέβαλε πρόταση για τον προϋπολογισμό του 2016 και βεβαίως είναι σαφές ότι Θέλουμε να υπάρξει χρηματοδότηση και των ζητημάτων που απασχολούν εμά ω Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη. Και συμφωνούμε όλοι, φαντάζομαι, ότι η Επιτροπή μας μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο θέμα αυτό. Τώρα, για τη διαδικασία του προϋπολογισμού είναι σημαντικό να ε, έρθουμε σε συνεννόηση με τον Γενικό Εισηγητή για τον προϋπολογισμό που είναι ο συνάδελφος Μανουέλ Φερνάντες. Χαίρομαι που βρίσκεται εδώ μαζί μας για να μας ενημερώσει ε, για τα θέματα που έχει θέσει αυτός ως πιο σημαντικά σχετικά με τον προϋπολισμό του 2016. Σας καλωσορίζω λοιπόν και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ είμαι ικανοποιημένος που είμαι ενώπιον της Επιτροπής σας. Έρχομαι κυρίως για να ακούσω τις δικές σας συμβουλές και ιδέες για να φτιάξουμε τον καλύτερο δυνατό προϋπολογισμό. Με βάση τα όρια βέβαια που πάντα διέπουν τους προπολογισμούς. Ψηφίσαμε τις κατευθυντηρίες ε, γραμμές 11 Μαρτίου 2015 με θέμα απασχόληση, επιχειρήσεις και κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρηματικότητα και επιχειρηματικό πνεύμα στο μυαλό μας. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να προωθήσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εξασφαλίζοντας την εσωτερική ε, αλληλεγγύη και είναι σημαντικό θέμα εδώ η εμπορική πολιτική. Ε, σε τα περισσότερα κατημέλη η πολιτική συνοχή σήμερα έχει διαφορετική, διαφορετικό ρόλο. Ε, συνεισφέρει στην έρευνα, στην έξυπνη ανάπτυξη. Ε, Επίση η εξωτερική αλληλεγγύη είναι σημαντική, είναι προτεραιότητα. Ε, η ασφάλεια όμως, η μετανάστευση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ξεχάσει τι συμβαίνει γύρω της παρά το γεγονός ότι συχνά ξεχνάμε ότι είμαστε οι μεγαλύτεροι δωρητές στον κόσμο βοήθειας. Ξεκινάμε από την αρχή ότι το Συμβούλιο και η Κομισιόν θα σεβαστούν τις ε, δεσμεύσεις τους. Δηλαδή το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο θα εξασφαλίσουν την ευελιξία που υπάρχει στον δημοσιο... πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τα περιθώρια για ε, απρόβλεπτα πράγματα. Το να σεβαστούμε λοιπόν τις δεσμεύσεις είναι να πληρώσουμε και τα χρέη. Είναι περίεργο που μιλάμε για πληρωμές που είναι λογική συνέπεια των δεσμεύσεων. Εδώ είχαμε μια συμφωνία με το Συμβούλιο και την Κομισιόν, ούτω ώστε οι καθυστερημένες πληρωμές του το 2016 να φτάσουν στο επίπεδο των 2 δισεκατομμυρίων. Η Κομισιόν έκανε την πρότασή της για το τελευταίο, στις 27 μάλλον Μαΐου, ε, για το προσχέδιο. Θα έχει μια ιδιαιτερότητα αυτό το προσχέδιο, γιατί η συμφωνία που είχαμε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Διασωτικών Επενδύσεων, το σχέδιο Γιούνκερ όπως λέγεται, η συμφωνία έχει ε, επίπτωση στα περιθώρια και μειώσαμε τις περικοπές του ορίζοντα 2020 και του Connecting Europe Facility αντί για 6 δις, 5 δις. Κερδίσαμε δηλαδή 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Για το χρονοδιάγραμμα, 23 Ιουνίου υιοθετούμε την έκθεση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών για την εντολή του τριμερούς διαλόγου που θα ε, ψηφιστεί α, τον Σεπτέμβριο. Ε, θα καταθέσουν οι βουλευτές μέσα ε, ε, Σεπτεμβρίου θα υιοθετηθεί η έκθεση για να υιοθετηθεί το ψήφισμα τον Οκτώβριο. Ε, θα ψηφίσουμε τις ε, τροπολογίες 12-13 Οκτωβρίου. Θα ψηφίσουμε για το ψήφισμα 28 Οκτωβρίου. Θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια 29 Οκτωβρίου και 18 Νοεμβρίου έχουμε την συνδιαλλαγή. Για το σχέδιο προπολογισμού το οποίο παρουσιάστηκε στις 27 Μαΐου για την μακροοικονομική βοήθεια. Για τις δεσμεύσεις 2,2% αύξηση για τις πληρωμές 7,3%. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία συνδέονται με αυτή την επιτροπή, με την δική επιτροπή, αλλά είναι το Ταμείο Εγγύσεων για τις εξωτερικές δράσεις σε επίπεδο δεσμεύσεων και πληρωμό 78% ε, έχουμε αύξηση. Για το εργαλείο εταιρική σχέσης έχουμε 6% στις δεσμεύσεις και 15,6% στις πληρωμές. στα πλαίσια της εσωτερικοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπάρχουν προγράμματα τα οποία είναι σημαντικά, αλλά και τα διαφορετικά ταμεία και τα επιχειρηματικά επιχειρηματικά προγράμματα σε κάθε χώρα είναι πολύ σημαντικά για το στόχο αυτό. Σας ευχαριστώ και ξέρω ότι στην Επιτροπή έχετε εμπειρογνώμονες εδώ, επαΐοντες για τα θέματα του προϋπολογισμού. που μπορούν να θέσουν τις προτεραιότητές σας και να τις, ε, να τις προτάξουν δηλαδή στην Επιτροπή Προϋπολογισμών για να λεφθούν υπόψη. Ευχαριστώ συνάδελφε Φερνάντες. Ναι, πράγματι. Τα έχουμε αυτά εδώ στην Επιτροπή Τα Δηλαδή έχουμε και εμείς ε, τις δυνατότητες να επιβάλλουμε κάποιες προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό. Και θα ήθελα να δώσω τον λόγο τώρα στον εισηγητή μας, τον κύριο Μπέγκε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ εισηγητά, αγαπητοί συνάδελφοι. Σε κοινή του συνεδρίαση σήμερα το βράδυ η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και Προϋπολογισμών ε, θα καταλήξουν σε συμφωνία και δεν ήταν καθόλου εύκολο. Η Κομισιόν επέλεξε τον ε, απλούστερο δρόμο όπως ομολόγησε και ήρθε σε συμφωνία με το Συμβούλιο. το Συμβούλιο. Άρα η αφιτηρία για το Κοινοβούλιο ήταν πολύ δύσκολη να σώσει ό,τι δίποτε κι αν σώζεται και να υπερασπιστεί τον ευρωπαϊκό προπολογισμό όσο καλύτερα μπορούσε. Έχω ε, εμπειρία όσον αφορά τις ε, δύσκολες διαπραγματεύσεις, αλλά όταν μετά από 13 ώρες διαπραγματεύσεις στον πέμπτο κύκλο ε, διαπραγματεύσεων του τριμερούς διαλόγου το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να εκφράσω πραγματικά το σεβασμό μου και την αναγνώρισή μου προς τους διαπραγματευτές μας ακόμη και ε, για την ε, γεγονός ότι διασώθηκαν ορισμένα εμβληματικά έργα ε, και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το Connecting Europe και θεωρώ ότι πρόκειται και για μια προειδοποιητική ε, βολή προς την Κομισιόν ώστε να τονίσουμε ότι χρειάζεται πιο προσεκτική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά το θέμα 4, το Global Europe, φυσικά από την ε, σκοπιά της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα ζητήματα του Διεθνούς Εμπορίου δεν θα πρέπει να εντάσσονται μόνο στο πρόγραμμα εργασιών της, της ε, Κομισιόν και να αναφέρονται ρητορικά, αλλά να αντικατοπτρίζεται μια τέτοια κατεύθυνση και στους συγκεκριμένους αριθμούς. Και αυτό θα μας απασχολήσει όσον αφορά και τα συμπεράσματα του ε, ε, ελεγκτικού συνεδρίου όπου τέθηκαν και κάποια ερωτήματα. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ε, σημαντική και απτή αύξηση των κονδυλίων για το διεθνές εμπόριο που σχετίζεται και με την ε, αξιολόγηση της εφαρμογής αλλά και των αποτελεσμάτων ε, που επιφέρουν οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε μόλις στην αρχή των όσων θα έπρεπε να, προβλη... θα έπρεπε να προβλέπονται. Θα πρέπει κάθε φορά να διασφαλίζουμε ότι γνωρίζουμε και ενημερωνόμαστε για το ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Πριν από μια εβδομάδα στην κοινοβουλευτική συνέλευση συζητήθηκε και στο Γερολάτε και, στο, και στη, στη με το ΣΕΛΑΚ. Υπάρχει μια πλειάδα θετικών, καλών ε, πρωτοβουλειών και αυτό που συζητούμε και εμείς ε, στις διαπραγματεύσεις μας με την Ινδία και την Κίνα αποτελεί θέμα σημαντικότατο και ε, στην σύναψη συμφωνιών μας με την Λατινική Αμερική ε, και πώς ε, τα πλεονεκτήματα από τις συμφωνίες αυτές μπορούν να βγουν προς όφελος και των μικρομεσαίων μας επιχειρήσεων γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξασφαλίσουμε αυτό που χρειαζόμαστε, δηλαδή τα μέσα για την ε, ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων των μικρών μεσαίων επιχειρήσεων, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό και για τους ε, εμπορικούς μας ε, εταίρους. Και όλα αυτά βεβαίως θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται και με τον δέοντα τρόπο στον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την ε, σύντομη μεν εξαιρετικά περιεκτική δε περιγραφή της εργασίας της Επιτροπής για τον προϋπολογισμό και την προετοιμασία αυτού για το 2016. Ένα σύντομο ερώτημα το οποίο θα σας εκπλήξει ενδεχομένως γιατί δεν έχει καμία σχέση με κάποιο εμπορικό ζήτημα. Ωστόσο, μου ήρθε αυτό το ερώτημα όταν άκουσα τις αρχικές σας παρατηρήσεις και όταν σας άκουσα να μιλάτε για θέματα που συνδέονται με την ασφάλεια, με την νόμιμη και παράνομη μετανάστευση και το καθεξής. Σημαίνει ότι υπάρχουν σχέδια ή γίνονται απόπειρες στον προϋπολογισμό, τον νέο προϋπολογισμό να αλλάξουν κατεύθυνση οι πόροι ή να δοθούν περισσότεροι πόροι για την προστασία των εξωτερικών συνόρων και να βοηθηθούν οι χώρες οι οποίες ε, de facto αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα εξ ονόματος όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή η Ιταλία και η Ελλάδα, για να προστατεύσουν τα σύνορά τους από την παράτυπη μετανάστευση. Υπάρχουν ε, σχέδια για περισσότερους πόρους για το θέμα αυτό. Ε, υπάρχει κάτι σύγκριμα που μπορείτε να μας πείτε. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Σόλτς. Και εγώ ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετικά ε, περίπλοκη κατάσταση και να μας με το ε, Global Europe. Αναφέρθηκε το ζήτημα του χρέους. Σε ποιο βαθμό συνυπολογίζονται είτε υπέρ είτε κατά ποσά που προκύπτουν από τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Και πώς στο μέλλον θα μπορούσαμε με καλύτερο τρόπο να εξασφαλίσουμε την, αξιοποίηση, την καλύτερη αξιοποίηση των ίδιων πόρων για να μπορούμε να επηρεάσουμε καλύτερα και τις ε, διεθνείς εμπορικές σχέσεις. Επίσης, το Trade World θα μπορούσε να αποτελέσει στο μέλλον ένα εργαλείο για να δημιουργήσουμε εμείς έναν άλλον μηχανισμό προκειμένου να παρακολουθούμε τέτοια ζητήματα και προκειμένου να μπορούμε να δίνουμε απαντήσεις στους πολίτες των 28 κρατών μελών μας αλλά και απέναντι στις Στου εμπορικού μα εταίρου, στι τρίτες χώρες για να μπορούμε να έχουμε απαντήσει πώ αυτέ οι διεθνεί εμπορικέ συμφωνίε τελικά επηρεάζουν και τι είδου επιπτώσει έχουν στι κοινωνίε των ε, συμβαλόμενων χωρών. Ευχαριστώ. Να, θέσω και εγώ, να κάνω και εγώ μια παρατήρηση που αφορά κυρίω την Κομισιόν. Αφενό υπάρχει η κατάσταση όπου βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορες ε, διμερείς ε, διαπραγματεύσεις και ενδεχομένω στο μέλλον να προσθεθούν και διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες, Μεξικό, Τουρκία, την Ισία και ταυτόχρονα δεν έχουν αυξηθεί οι πόροι που έχουμε στην ε, διάθεσή μας. Μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές διεξάγονται με τον ορθό και με τον κατάλογο τρόπο χωρίς να αυξηθούν τα κονδύλια και οι πόροι που βρίσκονται στη διάθεση της DG εμπορίου. Δεύτερο θέμα. Αν θέλουμε να πάρουμε στα σοβαρά τη συζήτηση για τις πολιτικές προτεραιότητες, φυσικά στο μέλλον δεν θα μπορούμε να συζητούμε μόνο κάθε φορά τις νέες προτάσεις ή τα νέα θέματα που θα τίθενται επί τα αλλά θα πρέπει να συζητούμε και τον έλεγχο της εφαρμογής αυτών των συμφωνιών. Ο κ. Μπέγκερτ το υπονόησε ότι είναι απαραίτητο να παρακολουθείτε και η εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών και να εξασφαλίζεται η ορθή επιβολή, εφαρμογή αυτών των ε, συμφωνιών. Και αυτό βεβαίως απαιτεί πόρους. Και εμείς θέλουμε ξεκάθαρα να ε, ε, συνεχίσουμε την ε, παρακολούθηση και της επιβολής της εφαρμογής αυτών των συμφωνιών. Και ένα θέμα που σχετίζεται και με το επόμενο ζήτημα που θα συζητήσουμε για την προσχώρηση ε, στην εμπορική συμφωνία με το Περού και την Κολομβία. Θέλουμε βεβαίως να συνάπτονται τέτοιες εμπορικές συμφωνίες αλλά θα πρέπει να είναι ε, δυνατή και η παρακολούθηση τη εφαρμογής αυτών των συμφωνιών. Και βεβαίως ε, κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει και μελέτη επιπτώσεων σε έναν προϋπολογισμό προκειμένου να μπορούν να λαμβάνονται και διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση που εμφανίζονται ε, προβλήματα. Ο κ. Μπόγκερτ. Ναι, ε, δύο-τρία συμπληρωματικά πράγματα θα ήθελα να πω. Θεωρώ ότι το ζήτημα των αποκλεινικών θέσεων είναι σημαντικότατο θέμα ε, στο παρελθόν ε, η Κομισιόν ε, έχει επιμείνει ότι εκείνη γνωρίζει καλύτερα ποιες είναι οι ανάγκες στις διάφορες γενικές διευθύνσεις. Ο κύριος Λικάνεν κάποτε όμως Φιλανδός είχε κάνει μια διοικητική μεταρρύθμιση ε, στην ε, Κομισιόν και όταν η μεταρρύθμιση του κατέληξε σε καταστροφικά αποτελέσματα η Κομισιόν είχε πει ότι η αρχή του προϋπολογισμού δεν της είχε δώσει ε, τις κατάλληλες θέσεις και εμείς απαντήσαμε ότι δυστυχώς δεν είχατε ζητήσει, δεν είχατε υποβάλει ποτέ έτοιμα για επιπλέον θέσεις και αυτό το ζητήματα που σχετίζεται με το, με το διεθνές εμπόριο με την, στο θέμα της Eurolat είχαμε την ε, αξιολόγηση ενός συναδέλφου από την ε, Νικαράγουα ο οποίος είχε επεξεργαστεί το θέμα της εξέλιξης των εμπορικών σχέσεων με τη Λατινική Αμερική και είχε καταλήξει και σε ένα έγγραφο το οποίο ήταν καλύτερο τελικά όσον αφορά την αξιολόγηση αυτών των συμφωνιών και της εφαρμογής τους από εκείνο που είχαμε από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Οπότε, το ερώτημα που θέτουμε εμείς είναι είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Ε, μπορούν τελικά αυτά τα θέματα που έχουμε, στα οποία εμείς έχουμε επιμείνει είναι εφικτό να εφαρμόζονται και να πω και κάτι κάπως προκλητικά. Εντάξει, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ε, βρίσκεται εκτός προϋπολογισμού. Από την άλλη πλευρά όμως αν εξετάσει κανείς όλα αυτά τα θέματα και αν ε, δει κανείς τι συμβαίνει στον νότο της Ευρώπης, δεν πιστεύω ότι μια ουσιώδη συζήτηση γύρω από το πώς θα χειριστούμε ε, τα ε, αναπτυξιακά εργαλεία δεν μπορεί να αναβληθεί για την περίοδο μετά τα 2020. Το θέμα της, ε, του προσανατολισμού των έργων είναι σημαντικότερο και ε, θα πρέπει να μας απασχολήσει το θέμα πώς θα αξιοποιούνται τελικά τα δικά μας κονδύλια ώστε οι άνθρωποι επιτόπου να ωφελούνται από την πολιτική μας και να μην έχουμε κατάσταση όπου δίνουμε ένα ε, ευρώ αναπτυξιακή βοήθεια και τελικά εγκαταλείπουν τη χώρα αυτή 10 ευρώ από διάφορους άλλους διάβλους. Ε, πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει όλες τις πολιτικές μας να τις ε, ε, αναθεωρούμε κατά διαστήματα προκειμένου να συντάσσεται και να χαράσετε μια ορθή πολιτική και καλό θα ήταν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφραστεί επί του θέματος αυτού. Κύριε Μπέγκερτ, λέει ο Πρόεδρος, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε και θα το δούμε και σε σχέση με την στρατηγική για το διεθνές εμπόριο που θα υποβάλει, θα προτείνει η Κομισιόν, ε, ελπίζω στο άμεσο μέλλον, γιατί θα πρέπει να παρακολουθούμε από κοντά τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Το άλλο ζήτημα που σχετίζεται με τους σπόρους, ε, σίγουρα είναι ένα θέμα στο οποίο θα μας ε, απαντήσει ο κύριος ε, εκπρόσωπος της Κομισιόν, ο κύριος Πέτσεσέλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Φερναντές και τους λοιπούς για τα πολύ ενδιαφέροντα που είπαν σε μια προηγούμενη ζωή ήμουν εκπρόσωπος τύπου του Επιτρόπου Λικάνεν, αλλά δεν θα σχολιάσω κάτι που είπε ή ενδεχομένω δεν είπε παλαιότερα. Τώρα για το θέμα των πόρων που θέτεται. Και εσείς κύριε Πρόεδρε και ο κύριος Μπέργκερ έχετε υπογραμμίσει κάτι το πολύ σημαντικό καθώς προχωράει η εμπορική ατζέντα. Έχουμε μια πολύ βεβαρημένη εμπορική σχετική ατζέντα διαπραγμάτευσης και βλέπουμε κάποιο φως στην άκρη του τούνελ. Υπάρχει ένα κύμα υλοποίησης το οποίο θα σκάσει, θα φτάσει στην ακτή λίαν συντόμως και αν είμαστε αισιόδοξοι μπορεί αυτό να γίνει μέχρι τα τέλη της επόμενης χρονιάς. Να έχουμε εφαρμόσει έξι νέες συμφωνίες σε περισσότερες από 13 χώρες, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι στην Αφρική. Όλα αυτά θα απαιτήσουν πολύ εντατική, πλευρά από, από, πολύ εντατική δουλειά από πλευράς μας. Ε, οι διαπραγματεύσεις είναι καλές, το θέμα είναι πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά. Και τρίτον, κάτι το οποίο είπε και το ελεγκτικό συνέδριο πέρσι, είναι σημαντικό τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των πραγμάτων που προτείνει με βάση τα στοιχεία και όλα αυτά να τα συνδέσει με το πακέτο μέτρων για καλύτερη νομοθεσία και εμείς και άλλες υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσπαθήσουμε, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τους διαθέσιμους πόρους. Αν όμως θέλουμε το εμπόριο πραγματικά το διεθνές να συμβάλλει στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ε, πρέπει να αξιοποιήσουμε τους πόρους με τον ε, πιο αποτελεσματικό τρόπο ή δυνατόν. Και Γι' αυτό ενδεχομένως πρέπει να αποφασίσουμε για προτεραιότητες και ε, για το που θα δώσουμε έμφαση. Είμαι κάπως προσεκτικός ε, για, όταν ακούω ιδέες για νέες δομές, όπως μια δομή παρακολούθησης των διεθνών εξελίξεων στο εμπορικό τομέα, Trade Watch Structure. Είναι πράγματα που έχουμε ήδη με τον επικοδομητικό και διαρθρωμένο και δομημένο διάλογο με την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, ε, με τα κεφάλαια ε, για την αηφόρο ανάπτυξη που αποτελούν μέρος των εμπορικών συμφωνιών. Αν έπρεπε να διαλέξουμε θα δίναμε μεγαλύτερη έμφαση στην επικοινωνία, στο να είναι όλοι ενημερωμένοι και να εμπλέκονται όσο το περισσότερο στις συζητήσεις για τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Φαίνεται ότι η συζήτηση μονοπολεί ε, το TTIP ε, τον τελευταίο χρόνο ή ενάμιση χρόνο και από πλευράς επικοινωνίας ε, θα ήταν καλύτερο να δώσουμε έμφαση εκεί και να δώσουμε προτεραιότητα στην επικοινωνία κυρίως και λιγότερο στο Trade Watch Structure. Σε κάθε περίπτωση με τον πεπερασμένο προϋπολογισμό εμείς υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να τον αξιοποιήσουμε και στην Γενική Διεύθυνση για το Εμπόριο και ε, για το ε, εργαλείο ε, σε σχέση με την ανατολική γειτονία. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αξιοποιήσουμε όλα τα δυνατά εργαλεία για την, στην, στις που έχουμε με τις τρίτες χώρες. Ευχαριστώ κύριος Φερναντές. Να σας υπενθυμίσω ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μικρός. Είναι το 1% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος ενώ στη ΣΥΠΑ είναι το 20% του ΑΕΠ, του εγχώριου ε, προϊόντος. Είναι όμως σημαντικός. Έχουμε 6% αυτού του προϋπολογισμού για τις διοικητικές δαπάνες, δηλαδή το 94% ε, του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού το έχουμε για τις επενδύσεις και αυτό το επαναλαμβάνω συνεχώς γιατί αυτό που λέω, λέει ο κ. Φερναντές, καταδεικνύει, αναδεικνύει πόσο προστιθέμενη αξία έχει ο προϋπολογισμός μας. Ο τίτλος 3, ε, ασφάλεια, είναι σαφέστατος. Εκεί έχουμε αύξηση των πόρων ή του ποσοστού αν θέλετε ε, για τα σύνορα και για τις χώρες. Από μνήμη σας λέω ότι για τη διαχείριση διαχείριση των συνόρων για την Ελλάδα πήγαμε στα 150 εκατομμύρια ευρώ από πολύ λιγότερα πριν, ενώ μέσα στον ίδιο τρίτο τίτλο θα αξιοποιήσουμε και θα φτάσουμε στα 124 εκατομμύρια ευρώ για το μέσο ε, ευελιξίας δεν έχουμε περιθώριο όμως και θα σας πω το εξή. Λέγεται ότι θα υπάρξει αύξηση, αύξηση, αύξηση. Όμως εγώ μιλώ για το σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θέλω να σας ευχηστήσω την προσοχή σε αυτό γιατί δεν έχει έρθει ακόμα η ανάγνωση αυτού του σχεδίου από πλευράς Συμβουλίου και το Συμβούλιο στην ανάγνωση που κάνει ενίοτε του σχεδίου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται και κάνει περικοπές ανεξήγητες το Συμβούλιο και πολύ συχνά αυτές οι περικοπές αντίκειται στις δεσμεύσει, στις πιστώσεις και στις δηλώσεις του Συμβουλίου για τις προτεραιότητες που υποτίθεται ότι έχει, μεταξύ άλλων. Έχουν συμβεί αυτά. Επομένως, να πούμε ότι εμείς αναλαμβάνουμε δέσμευση για τις συγκεκριμένες προτεραιότητες, θα περιμένουμε την ερμηνεία που θα δώσει το Συμβούλιο, τον τρόπο με τον οποίο θα αναγυγνώσει ε, το σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Συμβούλιο μάλλον θα προσπαθήσει να μειώσει τον προϋπολογισμό αυξάνοντας τα περιθώρια και να μην βάλει αρκετά χρήματα στο τραπέζι για τις πληρωμές, εξού και δημιουργείται το πρόβλημα με τις πληρωμές. Όμως, στον τίτλο 3, π.χ. στις δεσμεύσεις ε, έχουμε αύξηση 12,6% και στις πληρωμές 9,7% αντιστοίχως. Αναφέρομαι στο σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όταν επιμένω εδώ και επικαλούμε αυτά τα σημεία βλέπετε ε, πόση ελπίδα τρέφω και πόσο πολύ πιστεύω ή λίγο εντός εισαγωγικών ε, στην ανάγνωση που θα κάνει το Συμβούλιο. Στον τίτλο 4 για παράδειγμα βλέπουμε αύξηση των δεσμεύσεων 5,6% και στις, πληρώσει, στις πληρωμές 28,5%. Τι σημαίνει αυτό, ότι είναι σαφής η προτεραιότητα, φαίνεται και στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού, ότι είναι σαφέστατη η προτεραιότητα το όλο το θέμα του ασύλου, της μετανάστευσης των συνόρων και ούτω καθεξής. Ελπίζω το Συμβούλιο να έχει την ίδια προτεραιότητα. Ο Περέδη δείξε με την ανάγνωση που θα κάνει το Συμβούλιο. Είμαστε ένας, σε έναν προϋπολογισμό που δεν έχει αληθινούς ίδιους πόρους, αλλά είναι άλλη συζήτηση αυτή. Το 85% του προϋπολογισμού προέρχεται από το, ε, τους εθνικούς προϋπολογισμούς και αυτό είναι πρόβλημα. Θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η δουλειά έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει πραγματικά ίδιους πόρους. Τώρα στο θέμα του χρέους το οποίο δεν μπορούμε να έχουμε εδώ, γιατί αν διαβάσουμε τη συνθήκη δεν επιτρέπεται να έχουμε χρέος. Όμως, ε, Εάν υπάρχει κίνδυνος να διακινδυνεύσουν οι εξωτερικές συμφωνίες, λέω όχι. Βεβαίως όχι, δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Στα τέλη της χρονιάς θα έχουμε 20 δις καθυστερούμενες οφειλές πληρωμές, όμως το 2016 ελπίζουμε να, να πέσουμε στα 2 δις το μέσο όρο των ετών 2007 με 2013 δηλαδή. Και υπάρχει πρόβλημα με τα υπάρχει πρόβλημα με όσους ασκούν κριτική βεβαίως. Ε, βάσει της πολιτικής συνοχής έχουμε τον κανόνα νη 3 για την πολιτική συνοχή για την έρευνα, για την καινοτομία και το καθεξής και αυτό δημιουργεί πρόβλημα για τα ράλ. Τώρα, ε, συμφωνώ με την πρότασή σας, θα συνεχιστεί η δουλειά Υπάρχουν δυσκολίες στη διαπραγμάτευση, στη συζήτηση, όμως εμείς υπερασπιζόμαστε τις δικές σας απόψεις και όλα αυτά βρίσκονται στο σχέδιο έκθεσης που θα ψηφιστεί στις 23 Ιουνίου στην Επιτροπή για τον Προπολογισμό και στη συνέχεια θα πάει στην Ολομέλεια και ελπίζω ε, το Κοινοβούλιο να υιοθετήσει στεναρή θέση, αυτό το βλέπω σε όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, για να υπερασπιστεί την ανάπτυξη, την απασχόληση, την, την ασφάλεια και να βοηθήσει να λυθούν τα προβλήματα που έχουμε στα εξωτερικά μας σύνορα και κυρίως στη Μεσόγεια. Να, το Κοινοβούλιο να υιοθετήσει ε, σαφέστατη θέση για την εξωτερική και εσωτερική αλληλεγγύη και πάντοτε με σεβασμό στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Άλλωστε αυτό ζητούμε εμείς, να σεβαστεί κανείς το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν πάμε παραπέρα από αυτό το οποίο είναι εφικτό και να αξιοποιήσουμε τη συμβιβαστική λύση της ευελιξίας. Εμείς δεχθήκαμε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο να είναι σε πτώση γιατί είχε μπει εκεί στο πλαίσιο το θέμα της ευελιξίας. Και τώρα προκύπτει κάτι καινούριο για το οποίο δεν θέλει να γίνεται λόγο στο Συμβούλιο, αλλά εμείς το βάλαμε και το χρησιμοποιούμε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Ό,τι δηλαδή. Τα περιθώρια. Τα μη χρησιμοποιούμενα υπάρχουν. Άρα, στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αντίθετα με το προηγούμενο 2007-2013, τα μη χρησιμοποιημένα περιθώρια μιας οικονομικής χρήσης πάνε στην επόμενη χρήση ως ευρύτερα γενικά περιθώρια που μπορούν να διοχετευτούν σε συγκεκριμένη και ειδική πολιτική. Για λόγους λοιπόν αποτελεσματικότητας πρέπει να μπορούμε να αξιοποιούμε αυτά τα περιθώρια. Στον τίτλο 3 για παράδειγμα, για τον οποίο αναφερθήκαμε, από τη στιγμή που δεν υπάρχει περιθώριο, κινητοποιείται το μέσο της ευελιξίας εμείς όμως θέλουμε να υπάρχει περιθώριο στον τίτλο 3, π.χ. για τα πιλωτικά προγράμματα και για τι προπαρασκευαστικέ προπαρασκευαστικές δράσεις και θα υπερασπιστούμε αυτό το στόχο. Και αυτό που είναι απίστευτο είναι ότι ενίοτε έχω την αίσθηση ότι το Κοινοβούλιο υπερασπίζεται περισσότερο τις δεσμεύσεις, τις συμβαστικές λύσεις, την ανάπτυξη από ότι άλλοι. Και οι άλλοι θα έπρεπε να το κάνουν επίσης τόσο όσο και εμείς στο Κοινοβούλιο. Και οι άλλοι άλλα δηλώνουν και μετά έρχονται και πράττουν πράγματα που βρίσκονται σε αντίθεση με τις δηλώσεις τους και κυρίως με τις δηλώσεις που προκύπτουν μετά τις συνόδους κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Φερνάντες. Είναι πάντοτε πολύ συνεργαστικός ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή Προπολογισμών υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τις πολιτικές μας θέσεις στις ε, δύσκολες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Και αν εξετάσει κανείς ε, και το πόσες νέες ιδέες ε, έχει διαρκώς το Συμβούλιο για το τι πρέπει να χρηματοδοτεθεί, αλλά ταυτόχρονα και την έλλειψη πόρων για όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέρον το όλο θέμα. Εμείς ε, σε κάθε περίπτωση θα σας συνδράμουμε στο έργο σας και ελπίζουμε και σας ευχόμαστε να μπορέσετε να επιβάλλετε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις συγκεκριμένε διαπραγματεύσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Πρόταση του, την πρόταση του εισηγητή μας, του κυρίου Μπέγκερτ, θα τη συζητήσουμε στην τελευταία μας συνεδρίαση πριν από το καλοκαίρι που θα γίνει 13 και 14 Ιουλίου. Περνάμε στο θέμα 17. Την προσχώρηση του Εκουαδόρ στην εμπορική συμφωνία που έχει συναυθεί με την Κολομβία και το Περού. Να δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Σόλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε λίγες μέρες μετά την 8η Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΕΛΑΚ που ασχολήθηκε και με εμπορικά θέματα ή ασχολήθηκε κατά κύριο λόγο με εμπορικά θέματα θα πρότεινα να συζητήσουμε σήμερα την προτινόμενη προσχώρηση του Εκουαδόρ στην συμφωνία που έχει συναυτεί μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και ε, Κολομβίας ε, και Περού. Να σας ενημερώσω για το ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την προσχώρηση του Εκουαδόρ στη συμφωνία με, το, με την Κολομβία και το Περού. Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν, ε, οριστικοποιήθηκαν μάλλον συγγνώμη, τον Ιούλιο του 2014 και η συμφωνία ε, μονογράφηκε στις 12 Δεκεμβρίου του 2014 ενώ το κείμενο της συμφωνίας βρίσκεται στο στάδιο του ε, νομικού ελέγχου και της μετάφρασης και στη συνέχεια θα πρέπει να υπογραφεί και να κυρωθεί. Αν εξετάσουμε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, είναι σαφές ότι είναι μάλλον ε, απίθανο να οριστικοποιηθεί η όλη διαδικασία της κύρωσης πριν από το καλοκαίρι, παρά το γεγονός ότι έχει περάσει ήδη ένα, καλο, ένας ολόκληρος χρόνος και ε, προβλέπεται η θέση σε ισχύ στο τέλος του Ιουνίου. Στη συνέχεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν εξελιχθούν έτσι θετικά τα πράγματα το θα δώσει την σύμφωνη γνώμη του το 2016. Δεύτερον, να επισημάνω το γεγονός ότι παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλέον ε, ρήτρα GSP Plus για το Εκουαδόρ, ως συνομοθέτες από κοινού με το Συμβούλιο είχαμε συμφωνήσει να υπάρξει μια ε, προσωρινή ε, αναστολή των δασμών μετά την ε, οριστικοποίηση της συμφωνίας του 2014 και αυτή η αναστολή θα ισχύσει για δύο χρόνια έως ότου ολοκληρωθεί η δικασία κύρωσης έως ότου δηλαδή το Εκουαδόρ ολοκληρώσει και επισήμως την προσχώρησή του σε αυτή τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Κολομβίας και Περού. Πρόκειται δηλαδή για μια ε, αμοιβαία αναστολή των δασμών και απαιτεί και από εμά να, να λειτουργήσουμε με υπευθυνότητα όσον αφορά τη διαδικασία ε, κύρωσης οι ε, ε, η μη ασφαλείς μάλλον ε, ε, συνθήκες εργασίας οδηγούν σε οικονομικές απώλειες και αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Έχουμε να διαδραματίσουμε έναν σημαντικό ρόλο στο να προωθηθούν τα εργατικά δικαιώματα και τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Θα επιδιώξουμε την ε, περαιτέρω προώθηση και ε, ενίσχυση των ε, εργατικών προτύπων, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των συμφωνιών του ΟΗΕ, του ILO και τις ισχύουσες περιβαλλοντικές συμφωνίες σε όλη την παγκόσμια αλυσίδα τροφοδοσίας. Δεν είναι παράθεση από το πρόγραμμα της ΓΚΟΕ, αλλά Προέρχεται το κείμενο που σας διάβασα από την ε, ανακοίνωση που βγήκε έπειτα από τη συνεδρίαση των G7 φέτος τον Ιούνιο και αν, ακού, αν προσέξει κανείς ποιος συμμετέχει σε αυτόν τον μηχανισμό ε, θα ε, ε, λέγαμε ότι δεν είναι και ιδιαίτερα επικριτική όσον αφορά τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης είναι σημαντικό διότι οι συμμετέχοντες σε αυτήν την ε, σύνοδο κορυφής, τον G7, αναγνώρισαν την ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι τρίτων χωρών, δηλαδή των εμπορικών μας εταίρων και ιδιαίτερα απέναντι σε εμπορικούς εταίρους που δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ανάπτυξης από εμπορικής και οικονομικής άποψης όπως ε, είναι, ε, όπως στο επίπεδο δηλαδή που βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το λόγο δεν θα σας εκπλήξει το γεγονός ότι στο προτινόμενο ψήφισμα γίνεται αναφορά και στην ε, πτυχή της βιώσιμης και οικολογικής ανάπτυξης, διότι είναι σαφές ότι και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ευθύνη το εμπόριο να μην είναι μόνο ελεύθερο, αλλά να είναι και δίκαιο, ιδιαίτερα ε, για όλα τα μέρη που συμμετέχουν σε, αυτή, σε αυτές τις εμπορικές σχέσεις. Άρα αυτό δεν έχει μόνο ως αποτέλεσμα τη μείωση των δασμών, αλλά απαιτεί και συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων, για την, κατανάλωση, για την προστασία των καταναλωτών, για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών που συμμετέχουν στην σύναυση αυτού του είδους των εμπορικών συμφωνιών, αλλά απαιτεί και ε, μέτρα όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία δηλαδή των πολιτών, ε, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του Εκουαδόρ. Και γνώμη μου είναι ότι ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να εκφράσουμε με σαφήνεια μιας και ε, πρόκειται για μια ε, διαδικασία προσχώρησης ότι το Εκουαδόρ βρίσκεται σε μια θετική πορεία. Ε, οι δείκτες από την οικονομία του Εκουαδόρ είναι θετικοί, έχουν, αποτυπώνουν τις θετικές οικονομικές εξελίξεις που έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια στη συγκεκριμένη χώρα και αποδεικνύουν ότι, η, ε, ότι έχει υπάρξει μείωση σε σημαντικό βαθμό ε, της απόστασης που χωρίζει τα χαμηλά και τα υψηλά εισοδήματα. Ενώ φαίνεται ότι υπάρχει και μία ε, ενισχυόμενη μεσαία τάξη που είναι σημαντική και για την δημιουργία και την δραστηριοποίηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μεταξύ 2006 και 2014 η ανεργία μειώθηκε από 36% σε 22% ενώ μειώθηκε σημαντικότατα και ε, το ποσοστό πληθυσμού που ζει σε εθνικές ακραίας φτώχειας. Υπάρχουν δηλαδή θετικές τάσεις που είναι σαφείς και από αυτήν την άποψη είναι θετικό το γεγονός ότι η συγκεκριμένη χώρα προσχωρεί στη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Περού και Κολομβίας και ε, εμείς δεν θα πρέπει από την πλευρά μας να υπονομεύσουμε αυτή τη θετική διαδικασία και αυτή τη θετική τάση που έχει διαγραφεί στη συγκεκριμένη χώρα. Αυτό σημαίνει ότι η προσχώρηση του Εκουαδόρ στην συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κολομβίας και Περού θα πρέπει να διασφαλίζει ότι το Εκουαδόρ δεν θα συμμετέχει στη συμφωνία αυτή από μειονεκτική θέση. Προσωπικά ήμουν μεταξύ εκείνων που υποστήριξαν την οικολογική και κοινωνική βιώσιμη ανάπτυξη στο Εκουαδόρ και γι' αυτόν τον λόγο θα ήθελα να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως είχε εκφραστεί στις 11 Δεκεμβρίου του 2012 όταν δώσαμε τη σύμφωνη γνώμη μας για την προσχώρηση του Εκουαδόρ στη συγκεκριμένη συμφωνία και τότε είχαμε ε, πει και είχαμε τονίσει ότι είχαμε καλέσει μάλλον ότι θα πρέπει τα άλλα δύο κράτη της συμφωνίας να ε, συντάξουν μια διαφανή αλλά πάνω απ' όλα δεσμευτική ε, σειρά μέτρων που θα σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία του ε, του περιβάλλοντος. Και μάλιστα οι δύο κυβερνήσεις του Περού και της Κολομβίας τότε είχαν παρουσιάσει σχέδια δράσης και μάλιστα είχαν ξεκινήσει και την εφαρμογή αυτών των σχεδίων και φέτος στην Επιτροπή μας είχαμε ασχοληθεί διεξοδικά και με την εφαρμογή των συγκεκριμένων οδικών χαρτών και θεωρώ ότι θα πρέπει και στο μέλλον να παρακολουθούμε την εφαρμογή αυτών των οδικών χαρτών διότι αποτελούν προϋπόθεση ή αποτέλεσαν προϋπόθεση για να δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την σύμφωνη γνώμη του για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Περού και Κολομβίας και πιστεύω ότι είναι ευθύνη μας να παρακολουθούμε από κοντά την εφαρμογή αυτών των συμφωνιών ε, για να γνωρίζουμε σε περίπτωση που έχουν υπάρξει παρεκκλήσει από την εφαρμογή αυτή τη συμφωνία. τι είδους επιπτώσει θα υπήρχαν και για το Εκουαδόρ. Το Εκουαδόρ υπέγραψε λοιπόν τη συγκεκριμένη συμφωνία και μάλιστα ε, ανέλαβε και συγκεκριμένες δύο δεσμεύσεις για τη μεταρρύθμιση του τρόπου λειτουργίας της οικονομίας του. Γνωρίζουμε ότι η χώρα βασίζεται ε, σε μεγάλο βαθμό και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το δολάριο. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και αυτό το συγκεκριμένο γεγονός. Και γι' αυτό τον λόγο θα ήθελα να σας ζητήσω στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αντικατοπτρίζονται αυτές οι τροποποιηθήσεις ε, οικονομικές συνθήκες και να τονίσουμε ότι παρόλα τα προβλήματα υπήρξαν θετικά βήματα από την πλευρά του Εκουαδόρ όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, των εργαζομένων, των αυτοχθόνων και όσον αφορά την στήριξη και την ενίσχυση του τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελεί σημαντικότατο στοιχείο για την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας της χώρας. Και ταυτόχρονα υπήρξαν και σημαντικότατα μέτρα για την εξασφάλιση των επενδυτών και για την, την ισοτίμηση των ε, ε, ξένων αλλά και των εχώριων επενδυτών επενδυτών. Εξακολουθούν να υπάρχουν ε, ακόμη ζητήματα ανοιχτά που σχετίζονται με τα εργασιακά δικαιώματα σε αυτή τη χώρα, παρά το γεγονός ότι έχει η χώρα κυρώσει και τα 8 πρότυπα του διεθνού, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτά τα πρότυπα έχουν ε, υλοποιηθεί όλα αυτά τα πρότυπα και στην πράξη. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στο πρότυπο 129 ή στο πρότυπο 87. Και το θέμα αυτό το έχουμε συζητήσει και με εκπροσώπους του ΑΕΛΟ για να γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η κατάσταση στη χώρα. Θα ήθελα δηλαδή να αντικατοπτρίζονται στο ψήφισμα και οι εμπειρίες που έχουν συλλέξει αυτές οι ομάδες παρακολούθησης. Και για να τελειώσω, το Εκουαδόρ είναι ε, μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη βιοπικιλότητα, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ε, και αντίστοιχων ε, προβλημάτων που σχετίζονται με την βιοπικιλότητα. Άρα αυτό ε, μας θέτει και εμάς εν συγκεκριμένων ευθυνών και συγκεκριμένα για τη διατήρηση αυτής της βιοπικιλότητας. Για παράδειγμα, στο Εκουαδόρ υπάρχει ξεχωριστό Υπουργείο για την διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της χώρας. Γνωρίζετε το θέμα για Σούνη ITT, με το οποίο ασχολείται και το συγκεκριμένο Υπουργείο. Άρα εμείς θα πρέπει να εξετάσουμε πώς η προσχώρηση ε, σε αυτήν την Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου θα ε, διαφυλαχθεί και αυτή η κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση για την ε, κοινωνική και περιβαλλοντική ισορροπία. Δηλαδή θα πρέπει να διασφαλίσουμε να μην υπάρξει περαιτέρω διάευρωση του εδάφους, να μην υπάρξει μόλυνση των υδάτινων πόρων, να υπάρχουν στο ψήφισμα δεσμευτικοί στόχοι ε, όσον αφορά τη δραστηριοποίηση Ευρωπαίων επενδυτών στο Εκουαδόρ προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη αυτή η ιδιαίτερα περίπλοκη κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η Κομισιόν θα πρέπει να ενισχύσουν την, τις προσπάθειες και να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της κυβέρνησης του Εκουαδόρ για να ε, συνεχίστη η εφαρμογή σχετικών ε, προγραμμάτων στη χώρα που σχετίζονται και με την διαφύλαξη της περιοχής του Αμαζονίου. Από αυτή την άποψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω ε, ως δεσμευτική μάλιστα υποχρέωση την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Και τέλος όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα που έχει καταρτιστεί το χρονοδιάγραμμα είναι το εξής. Το σχέδιο ψηφίσματος θα το συζητήσουμε στις 13-14 Ιουλίου και στη συνέχεια έως τις 17 Ιουλίου, αν εγκριθεί το ψήφισμα, θα έχουμε χρόνο για την υποβολή τροπολογιών και στη συνέχεια στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου θα μπορέσουμε να συζητήσουμε σε δεύτερη ανάγνωση ε, το ψήφισμα αυτό, να συζητήσουμε τις τροπολογίες ώστε στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην υπερψήφιση του ψηφίσματος, όπως είπα στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και βεβαίως είμαι ε, πρόθυμος να ακούσω και τις απόψεις των ε, συναδέλφων. Ευχαριστώ Χέλμουντ. Σε ευχαριστούμε για την παρουσίαση της ε, ισχύουση κατάστασης. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον μόνιμο ισογητή μας για, τον, ε, για την Κολομβία και το Περού. Ο λόγος στον κύριο Φίσας. Ευχαριστώ πρόεδρε. ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Σόλτς για αυτή την πλήρη παρουσίαση και για όλη τη δουλειά που γίνεται για την ε, ένταξη του Εκουαδόρ σε αυτή την εμπορική συμφωνία που ισχύει αυτή τη στιγμή με την Κολομβία και το Περού. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι αυτή η συμφωνία, εμπορική συμφωνία, έγινε τον Ιούλιο του 2014 και προέβλεπε και το Εκουαδόρ και τη Βολιβία ως μέλη του. Αλλά οι χώρες αυτές αποφάσισαν να μην το υπογράψουν. Εν συνεχεία το Εκουαδόρ ε, σκέφτηκε ότι ήταν ενδιαφέρουσα αυτή η συμφωνία και αποφάσισε να ενταχθεί στην εμπορική συμφωνία με τις χώρες των Άνδεων. Θα ήθελα να πω ότι όταν κάποιες πολιτικές ομάδες λένε, λένε ότι εμείς υποχρεώνουμε κάποιες χώρες του τρίτου κόσμου να υπογράψουν ε, συμφωνίες, αυτό δεν ισχύει. Και αυτή είναι η απόδειξη. Ότι το Εκουαδόρ, επειδή είδε κάτι καλό στη συμφωνία, την εμπορική αυτή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζήτησε μόνο του να ενταχθεί σε αυτή τη συμφωνία. Κανένα δεν υποχρέωσε το Εκουαδόρ να ενταχθεί. Ήταν δύσκολε οι διαπραγματεύσεις. Όλοι ξέρουμε ότι το Εκουαδόρ είχε τη μονομερή, α, μονομερής α, προτιμήσεις. Ε, τελείωσε ο νόμος στις 31 Δεκεμβρίου του 2014. Ε, ήταν δύσκολο αυτό λοιπόν για τις επιχειρήσεις του Εκουαδόρ που μετά την λήξη συμφωνίας άρχισαν να ψηλώνουν ψηλούς δασμούς. Για γενικευμένες προτιμήσεις. Υπήρχε δυνατότητα λοιπόν προσωρινά να ενταχθεί το Εκουαδόρ ούτως ώστε να μην πληρώνει αυτούς τους δασμούς. Χαίρομαι λοιπόν που το πράγμα πάει ακόμα πιο μακριά, προχωράει και που μπορεί να εγκριθεί το συντομότερο δυνατόν. Σε ό,τι αφορά την ε, διαβόητη, τον διαβόητο οδικό χάρτη. Αυτά, αυτοί οι οδικοί χάρτες δεν μας αρέσουν πάρα πολύ. Δεν υπάρχουν σε πολλές άλλες εμπορικές συμφωνίες, αλλά ούτε θα αντιταχθούμε. Γιατί την έχει αυτή τη στιγμή η Κολομβία και το Περού. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτήν την περίπτωση, γιατί η ένταξη του Εκουαδόρ δεν σημαίνει ότι γίνεται αυτό που γίνεται ακριβώς στην Κολομβία και στο Περού. Κάθε χώρα έχει τις δικές της συνθήκες. Δεν είναι οι ίδιες οι συνθήκες ε, στο Εκουαδόρ. Δεν διαφέρουν ε, με το Περού, με το Περού και της Κολομβίας. Ακόμα και της Κολομβίας με το Περού μεταξύ τους διαφέρουν. Νομίζω ότι αυτό σημείο θα πρέπει να το ψάξουμε. Η κυβέρνηση του Εκουαδόρ δεν ήταν πολύ ευνοϊκή να της επιβληθεί ένας οδικός χάρτης γιατί θεωρούσαν ότι ε, έχουν διαφορετικές συνθήκες αυτή η χώρα από τις άλλες χώρες. Από την άλλη μας επιτρέπει και μια σύγκριση, επομένως είναι ένα θέμα που πρέπει να το μελετήσουμε με μεγάλη προσοχή αυτό το δικού χάρτη. Ε, εμείς είμαστε υπέρ της ένταξης από την άλλη του Εκουαδόρ στη συνθήκη και ελπίζουμε οι διαπραγματεύσεις να γίνουν, όπως είπε και ο εισηγητής, χωρίς ε, περαιτέρω εμπόδια και το συντομότερο δυνατόν, να, οι διαδικασίες δηλαδή να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν και να μπορέσουμε ε, να εντάξουμε το Εκουαδόρ στην ε, εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι πολύ ευνοϊκό αυτό για, για τις επιχειρήσεις του Εκουαδόρ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως ο εισηγητής να είναι σίγουρος ότι έχει την εμπιστοσύνη μου και τη συνεργασία μου ε, και τη δική μου και της ε, πολιτικής μου ομάδας. Ευχαριστώ θερμά. Κυρία Ευχαριστώ. Επαναλαμβάνουμε τα θέματα του οδικού χάρτη. Είναι θέμα συνέπειας στις σχέσεις μας με την κοινότητα των Άνδεων. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε στο Κοινοβούλιο το 2012 μιλούσε για τις χώρες της ε, κοινότητας των Άνδων και δεν μιλούσε ρητά για την Κολομβία και το Περού ε, που ήταν όμως οι χώρες που υπέγραψαν τη συμφωνία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να συνεργαστούμε με τις αρχές του Εκουαδόρ για να αναπτύξουμε ένα οδικό χάρτη που να καλύπτει και το Εκουαδόρ. Υπάρχει μάλιστα η ευκαιρία σε αυτό το οδικό χάρτη για τις αρχές του Εκουαδόρ αν θέλουν να ασχοληθούν Υπάρχουν κάποια θέματα που δημιουργούν ανησυχίες. Υπήρξαν επισκέψεις ε, με τεχνικές αποστολές και υποβολές και μάλλον και ε, επιτροπές εμπειρογνωμόνων για τα δικαιο... τις συλλογικές συμβάσεις και διάφορα άλλα θέματα. Είναι σημαντικό να συζητήσουμε για τα θέματα ανησυχίας με τις αρχές του Εκουαδόρ και δεν θέλαμε να έχουμε τρεις ε, χώρες ε, εταίρους που έχουν υπογράψει την ίδια συμφωνία και οι δύο έχουν ε, υποβληθεί σε οδικό χάρτη, ενώ η τρίτη θα λέει όχι, καλύτερα είναι να, μην έχουμε εμεί οδικό χάρτη. Νομίζω ότι είναι σωστό να έχουμε ίδια προσέγγιση και στι τρει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς στην ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών ήμασταν υπέρ οποιασδήποτε συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου γενικότερα και τη συγκεκριμένη ειδικότερα με την Κολομβία και το Περού. Καλωσορίζουμε την προσχώρηση του Ισημερινού σε αυτή την ε, εμπορική συμφωνία, σε αυτές τις εμπορικές, εμπορικές ρυθμίσεις και κυρίως για τρεις λόγους. Πρώτον, διότι διασφαλίζεται η πρόσβαση στις αγορές. Δεύτερον, θα δημιουργήσει ένα σταθερό και παραγωγικό περιβάλλον. Και τρίτον, θα προωθήσει και θα διαφοροποιήσει το εμπόριο εκατέρωθεν. Και φυσικά στηρίζουμε αυτό το προσωρινό, να το χαρακτηρίσω, μέτρο του ESP Plus κανονισμού βάσει αυτής της συμφωνίας. Ε, το οποίο και θα εφαρμοστεί πλήρως. Θα ήθελα να τονίσω τα ενδυνάμει ωφέλη και ευκαιρίες που απορρέουν από τη συνθήκη. Όμως, δεν είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τα προαπαιτούμενα για δεσμευτικό οδικό χάρτη για κάτι τέτοιο για το οποίο έχουμε ήδη εγείρει αντιρρήσεις για την περίπτωση της Κολομβίας και του Περού. Άρα ούτε στον Ισημερινό ε, θα το ε, δεχθούμε και θα δεχθούμε πίεση από πλευράς ε, κυβέρνησης Κορία για θέματα περιβαλλοντικής εργατικής νομοθεσίας κτλ. Ε, κυβέρνηση του Εκουαδόρ, με συγχωρείτε. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε την κυβέρνηση του σημερινού και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τα περιβαλλοντικά πρότυπα και, και, και για την αγορά εργασίας μπορούμε να βοηθήσουμε, μπορούμε να ενθαρρύνουμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούν να τεθούν νέες κόκκινες γραμμές για τα θέματα αυτά που θα αποτελέσουν κόλλημα στις εμπορικές μας σχέσεις. Με αυτή την εξαίρεση λοιπόν στηρίζουμε τη συμφωνία, διακείμεθα ευμενός και θετικός και ελπίζουμε να είναι θετική απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Η κυρία Κέλλερ. I'm very sorry that I have to miss most of this back due to the voting in another committee. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Ε, ήρθα καθυστερημένα και, δεν, γι' αυτό δεν σας άκουσα. Η πράσινη η ομάδα μου δεν είναι υπέρ της α, ε, συμφωνίας. Δεν ήταν υπέρ της συμφωνίας αρχικά για το Περού και την Κολομβία ε, και είχαμε επιχειρήματα τα οποία δεν άλλαξαν. Τώρα μπαίνει και το Εκουαδόρ Θέλουμε βεβαίω δίκαιο εμπόριο, αλλά δεν πιστεύουμε ότι ο τρόπος που συνάπτουμε εμπορικές συμφωνίες πληρώνει τις προϋποθέσεις ε, δικαιοσύνης ας πούμε και αμοιβέ ωφέλεια. Για το Εκουαδόρ τώρα. Να ρωτήσω την Κομισιόν. Το θέμα της μπανάνας και των τιμών της μπανάνας πώς έχει αντιμετωπιστεί. Δεν ξέρω αν είναι στα των συζητήσεων μα. Γιατί ίσως θα υπάρξει πρόβλημα για τους παραγωγούς μπανάνα στο Εκουαδόρ αν ε, τους ε, επιβάλλουμε τις ίδιε ψήφου ε, δασμού με τους παραγωγούς του Περού και της Κολομβίας. Πώς θα αντιμετωπιστούμε, αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα και υπάρχουν αντιρρήσει από την εκουαδοριακή πλευρά για το θέμα τη μπανάνα, για το θέμα τη γαρίδα Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό το Εκουαδόρ, που είναι φτωχή χώρα, να μπορέσει να προστατεύσει τις βιομηχανίες που μόλις αρχίζουν να ξεμητίζουν. Θέλω να ρωτήσω επίσης την Κομισιόν με ποιο τρόπο η αναθεώρηση της του εγχειριδίου για την βιωσιμότητα του εμπορίου θα επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις, αν τις επηρεάσει, και για τον οδικό χάρτη πιστεύω ότι έχει κάποια όρια ο οδικός χάρτης. Ενώ αυτό που θέλουμε είναι ένα δεσμευτικό κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό το έχουν κάνει διάφορες χώρες και νομίζω ότι αυτό θα ήταν ο σωστό τρόπο να προχωρήσουμε. Δεν νομίζουμε ότι ο δικό χάρτης μας οδηγεί κάπου. Και ειδικά ο δικός χάρτης της Κολομβίας και του Περού που λέει αυτά, αυτά που λέει. Αν είχαμε ένα κοινό δικό χάρτη, τουλάχιστον να ήταν δεσμευτικό. Αλλά το βασικό είναι να υπάρχει ένα δεσμευτικό κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω εκεί στο πίσω μέρος της ε, αίθουσα την ε, διάδοχο του Γιώργ Λάιχτριτ που έγινε υπουργός στη Στηρία, στην, Ευ... στην Αυστρία, υπουργό συγκοινωνιών και η συνάδελφος ήρθε και μάλλον προσπαθεί να συνηθίσει και να εξοικειωθεί ε, με τις εργασίες μας και το χώρο. Το ζήτημα της, ε, του, του χειρισμού του οδικού χάρτη είναι σημαντικό. Υπάρχει ένα μοντέλο στη βάση των όσων κάναμε με την ε, Κολομβία και του Περού και στη βάση των ε, εμπειρών που συλλέξαμε θα πρέπει βεβαίως να βελτιώσουμε, ενδεχομένως να υποστηρίξουμε και περισσότερο δυνατότητες που υπάρχουν, ε, ιδιαίτερα όσον αφορά το εμπόριο λουλουδιών και μπανάνας με το Εκουαδόρ νομίζω ότι υπάρχουν δυνατότητες στήριξης του δίκαιου εμπορίου και ε, έχοντας υπόψη μου και το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα που διεξήχθη με, το, με την Κολομβία θεωρώ ότι είναι μια διαδικασία που θα μπορούσε να μεταφερθεί και στην περίπτωση του Εκουαδόρ. Την απέτηση δηλαδή να ε, λαμβάνονται μέτρα Βεβαίως το ότι υποστηρίζουμε την προσχώρηση είναι αναμφισβήτηση, αναμφισβήτητο και τα πλεονεκτήματα από μια τέτοια συμφωνία είναι προφανή, γι' αυτό θα πρέπει να οργανώσουμε με τέτοιο τρόπο τη μετάβαση ώστε να υπάρξουν ωφέλη και για την οικονομία και για την ε, κοινωνία για τις μπανάνες είχαμε κάποια προβλήματα και με τις ποσοστώσεις της Κολομβίας και η στάση της Κομισιόν δεν ήταν και πολύ σωστή σε εκείνο το θέμα. Το ερώτημά μας λοιπόν είναι ποια είναι η θέση τώρα της Κομισιόν. Νομίζω ότι ο εκπρόσωπος της Κομισιόν τα έχει συγκεντρώσει και θα έχει την ευκαιρία να μας απαντήσει σε όλα αυτά η πρόσωπος της Κομισιόν, η κυρία Κιόνικ. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσω από την αρχή, όπως είπε ο εισηγητής ο κύριος Σόλτς. Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο του 2014 και το πρωτόκολλο προσχώρησης υπογράφηκε από την Επίτροπο Μάλστρομ και τους Υπουργούς το Δεκέμβριο του 2014. Έκτοτε δύο τι να συμβαίνουν. Πρώτον μεταφράζεται σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και περιμένουμε την τελική επιβεβαίωση του συμπεφωνηθέντος κειμένου. Παράλληλα, ε, οι άλλες διαβουλεύσεις έχουμε ξεκινήσει με την Κολομβία και το Περού για τη συμφωνία τους για την προσχώρηση του Ισημερινού στη συγκεκριμένη εμπορική συμφωνία. Είναι τρέχουσα η διαβούλευση με αυτές τις δύο χώρες και θα ολοκληρωθεί πριν το τέλος του καλοκαιριού. Χρειάζεται περαιτέρω ε, χρόνος λόγω εσωτερικών συζητήσεων μέσα σε αυτές τις δύο χώρες και σε βασικές γραμμές η Κολομβία και το Περού εξέφρασαν το εξή. Είπαν ότι οι δικέ του ανησυχίες δεν έχουν να κάνουν με την προτινόμενη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με το τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στι σχέσει μεταξύ των τριών χωρών, στι υφιστάμενες συμφωνίε που έχουν οι τρει χώρε μεταξύ του. Και το συζητούμε αυτό και ελπίζουμε να βρεθεί λύση το συντομότερο δυνατό αυτή τη στιγμή. Επίσης έχουμε την Εμπορική Επιτροπή η οποία εξελίσσεται, λειτουργεί. Ε, την ε, Παρασκευή αυτή θα συνεδριάσει και έχουμε και την Υποεπιτροπή για το εμπόριο και την αεφόρο ανάπτυξη που συνδέεται με τα κεφάλαια αυτά που είναι υποσυζήτηση. Δεν ξέρω ποια θα είναι η έκβαση εκεί και τα δύο προφανώς θα συζητηθούν οι διατάξεις και οι δυνατότητες για την υπογραφή της συμφωνίας και η παρακολούθηση ε, του κεφαλαίου για την αηφόρο εμπορική ανάπτυξη. Τώρα, ως προς το πρωτοκόλλο αυτό καθεαυτό, προφανώς εναπόκειται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άπαξ και έχουμε τη συμφωνία με την Κολομβία και το Περού να εξετάσουμε αυτή την απόφαση. Θεωρούμε ότι θα έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας να εξετάσουμε το πρωτόκολλο, ένα πρωτόκολλο. Ο εισηγητής έχει ξεκινήσει τη συζήτηση και αυτό είναι εξαιρετικά θετικό. Δεν ξέρουμε πόσο γρήγορα θα είμαστε σε θέση να σας φέρουμε την οριστικοποιημένη τελική συμφωνία. Και ως προς τα ωφέλη της συμφωνίας, και νομίζω ότι ε, λίγα μελή το σχολίασαν αυτό της Επιτροπής σας, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή κάνουμε μια μελέτη για τον αντίκτυπο της συμφωνίας με τον Ισημερινό, με το Εκουαδόρ δηλαδή. Δεν έχει αυτό ολοκληρωθεί. Θα ολοκληρωθεί λίγο πριν το καλοκαίρι η απάντηση των δύο άλλων χωρών και άρα στις αρχές του φθινοπόρου θα ολοκληρωθεί η μελέτη αυτή από πλευράς μας ε, κατ' επέκταση. Το GSP-SYN ε, εποφελείται από από τη συμφωνία με τον, με τον Ισημερινό και έχουμε ετησίως εξοικονόμηση 200 ε, εκατομμυρίων ευρώ από πλευράς δασμών και έτσι προστατεύονται και οι εξαγωγές του Ισημερινού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι σημαντικό και για τον Ισημερινό αλλά και για μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Αυτά λοιπόν η εμπορική συμφωνία έχει επιπρόσθετα ωφέλη για τις μπανάνες προφανώς. Όπως σχολίασαν και ορισμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι μια συμφωνία την οποία επιθυμεί ο Σημερινός, όχι μόνο για το GSP, αλλά και για τη συνοχή στην ε, εκεί περιοχή και για τις υφιστάμενες ε, εμπορικές συμφωνίες θα τους βοηθήσει να προσελκύσουν FTI από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς από την πλευρά μας μας συμφέρει γιατί έχουμε σταθερότητα στο πλαίσιο. Τώρα, δύο λόγια για το κεφάλαιο εμπορίου και αηφόρου ανάπτυξης. Είναι βασικό για όλες τις συμφωνίες μας στη Λατινική Αμερική. Ο Ισημερινός έχει ήδη συμφωνήσει να προσυπογράψει τις διατάξεις όλες του κεφαλαίου για την αηφόρο εμπορική ανάπτυξη. Ωστόσο, εξέφρασε ανάγκη για ευελιξία στις διαπραγματεύσεις και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το ερμηνεύσουμε με τη θετική του σκοπιά. Δείχνει βούληση από τον Ισημερινό να είναι παρόν σε αυτό το τομέα και να αναλάβει δεσμεύσεις και αυτή η ανάληψη δέσμευσης είναι σημαντική, καθοριστική για να τεθεί σε ισχύ και να εφαρμοστεί η εκάστοτε διάταξη. Ε, ούτως ή η επιτυχία εξαρτάται από τη συνεργασία με τις χώρες με τις οποίες έχουμε συμφωνία. Η δήλωση του Ισημερινού δείχνει πόσο σημαντική είναι για αυτούς η περιβαλλοντική προστασία, τα εργατικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών. Και με την προσχώρηση του Ισημερινού στη συμφωνία θα βοηθηθούμε για να εντοπίσουμε μια κοινή ημερήσια διάταξη και για αυτά τα ζητήματα. Επιπρόσθετα, η συνεισφορά της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών θα είναι εξαιρετικά σημαντική και, και εκεί περιμένουμε θετική συνεισφορά του ησημερινού. Και τέλος, για το κεφάλαιο της εμπορικής αηφόρου ανάπτυξης, της αηφόρου εμπορικής ανάπτυξης. Δεν είναι αυτό το μόνο που μας απασχολεί για τη συμπλήρωση της εμπορικής συμφωνίας. Υπάρχουν και άλλα. Υπάρχει δέσμευση μεταξύ της δικής μας αντιπροσωπείας με τις αρχές και με την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών για όλα αυτά τα ζητήματα έχουμε αναλάβει τη δέσμευση. Τώρα έρχομαι στις ερωτήσεις που μου έχουν τεθεί. Ε, π.χ. για τις μπανάνες. Όπως ανέφερα, η συμφωνία καθρεφτίζει αυτό που έχουμε σε μεγάλο βαθμό με την Κολομβία και το Περού. Ε, διαφορά είναι μόνο τα στάδια εφαρμογής. Έχουμε τον κανονισμό για το μηχανισμό σταθεροποίησης της μπανάνας και τις εμπορικές δραστηριότητες αυτής. Ε, αυτό ε, αποτελεί μεγάλο μέρος της συμφωνίας με τον Ισημερινό. Δεύτερο ερώτημα για την αναθεώρηση του εχειριδίου για την ε, αηφόρο εμπορική ανάπτυξη. Βεβαίω είναι κάτι που επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρηση αυτή. Έχει οριστικοποιηθεί. Θα τη λάβουμε υπόψη μα τον τρόπο με τον οποίο θα εξετάσουμε την αφαρμογή τη συμφωνία. Δεν έχει αλλάξει όμως η συμφωνία αυτή καθεαυτή από το εγχειρίδιο, το handbook, γιατί η συμφωνία είχε οριστικοποιηθεί πριν οριστικοποιηθεί η αναθεώρηση του εγχειριδίου του handbook για την αηφόρα εμπορική ανάπτυξη. Ωστόσο, είναι κάτι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί σφόδρα να αναπτύξει στο μέλλον, να ε, ενισχύσει, να διευρύνει αν θέλετε και διαφορετικές πτυχές θα, του εχειριδίου για την εφόρο εμπορική ανάπτυξη, διάφορες διαστάσεις θα ληφθούν υπόψη στη συζήτηση για την στην υποεπιτροπή TSD. Κατά πόσο υπάρχουν διαφορετικές πρωτοβουλίες, κατά πόσο υπάρχουν μέτρα όλα αυτά θα τα δούμε, είμαστε ανοιχτοί να τα δούμε σε συνέργεια και συνεργασία με τους εταίρους μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά. Νομίζω ότι είναι σαφές πλέον και σε σχέση με το ψήφισμα ότι θα πρέπει να φωτίσουμε τα διάφορα δομικά στοιχεία που σχετίζονται με την εφαρμογή. Και μιας και το θέμα της εφαρμογής των συμφωνιών κινεί το ενδιαφέρον πολλών πλευρών. Θα έλεγα ότι όλοι αυτοί οι φορείς και όλες οι επιτροπές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα πρακτικά και στις συζητήσεις για το πώς η Ευρώπη ε, θα μπορούσε να ενισχύσει όλες αυτές τις πρωτοβουλίες θα πρέπει σε αυτήν τη διαδικασία να εμπλακεί όσο το δυνατόν περισσότερο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να προωθηθούν όλες αυτές οι διαδικασίες όσο το δυνατόν περισσότερο. Και αυτό ε, αφορά και το επερχόμενο ψήφισμα αλλά και τη μελλοντική, ε, τις μελλοντικές προσπάθειές μας για την ε, εφαρμογή των συμφοριών. Ο κύριος Σόλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το σημαντικότερο ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη προσοχή στην εφαρμογή αυτών των συμφωνιών και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρχουν ε, συγκεκριμένα δεσμευτικά νομικά βήματα που θα δεσμεύουν όλες τις πλευρές, όλα τα μέρη, στην, εμπροκειμένο το Εκουαδόρ, αλλά και την Κολομβία και το Περού, καθώς και τις άλλες δύο χώρες δηλαδή, αλλά θα πρέπει να ισχύουν οι δεσμεύσεις αυτές και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και από αυτή την άποψη θα πρέπει ένα τέτοιο συνοδευτικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ε, παραθέτει συγκεκριμένες υποχρεώσεις και για τους δικούς μας εμπλεκόμενους φορείς και να ορίζουμε τι ακριβώς θέλουμε να παρακολουθήσουμε και τι ακριβώς θέλουμε να ελέγξουμε όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας και να, να καταρτιστεί και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσεων και θα πρέπει αυτό να το έχουμε υπόψη μας, ιδιαίτερα και υπό το φως των συζητήσεων που είχαμε σήμερα το πρωί και χθες, δηλαδή το θέμα ε, ότι υπάρχει πλέον ένας πολυμερής, ε, ένα, μια πολυμερής συμφωνία εμπορική η οποία προβλέπει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις για όλα τα μέρη. Άρα θα πρέπει ως μέτρο σύγκρισης να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη οι καταστάσεις που ισχύουν και στις δύο πλευρές και θα πρέπει να ελέγχεται ε, συγκεκριμένα σε ποιους τομείς ελήφθησαν μέτρα στο Εκουαδόρ προκειμένου να δημιουργηθεί μια σύγχρονη οικονομία, πώς προστατεύτηκε το περιβάλλον, πώς προστατεύτηκαν οι αυτόχθονες πληθυσμοί, πώς τήρησε το, και με ποιον τρόπο τήρησε το ε, Εκουαδόρ τις διεθνείς του υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τι περαιτέρω δυνατότητες υπάρχουν ε, στους συγκεκριμένους τομείς στο μέλλον. Νομίζω ότι στο έργο μας της κατάρτισης του ψηφίσματος θα πρέπει όλα αυτά τα ζητήματα να ληφθούν ε, υπόψη και να συμπεριληφθούν και στο τελικό ψήφισμα. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Με μεγάλη αγωνία λοιπόν περιμένουμε την πρόταση το σχέδιο ψηφίσματος και όπως υπόθηκε και νωρίτερα, το σχέδιο αυτό θα συζητηθεί στην τελευταία μας συνεδρία πριν από το καλοκαίρι στις 13-14 ε, Ιουλίου. Περνάμε στο θέμα 18 ομάδες παρακολούθησης, εκτός από τη σύναψη δηλαδή συμφωνιών, θα πρέπει να υπάρχει και η παρακολούθηση αυτών των συμφωνιών και νομίζω ότι ε, αποτελεί πραγματικά παράδειγμα προς μίμηση αυτή η δημιουργία των ομάδων ε, παρακολούθησης ε, και Ακριβώς το ίδιο άλλωστε έχει ζητήσει πλέον και το, κον, το Κογκρέσο όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για το TTIP. Σε παγκόσμιο επίπεδο λοιπόν δημιουργούμε πλέον προδιαγραφές και πρότυπο. Λοιπόν, πρώτον, Μεξικό. Sorry. Ευχαριστώ. Συναντήθηκε στις 11 Μαΐου ε, η ομάδα παρακολούθησε για το Μεξικό επευκαιρία της επίσκεψης του Υπουργού Οικονομίας του Μεξικού που καλύπτει και θέματα εμπορίου όμως ε, στις Βρυξέλλες ήρθε για μια σειρά συνεδριάσεων με την Κομισιόν είδε την Επίτροπο Μάλστρομ και επαφών για να συζητήσει την προσπάθεια που είναι εξελίξει εδώ και δύο χρόνια μεταξύ Μεξικού και Κομισιόν για να εξυγχρονιστεί η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου που έχουμε με το Μεξικό. Με την ευκαιρία της παρουσίας του κάναμε μια ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων για το τι έχει συμβεί. Η συνάντηση ήταν ειδική, ιδιαίτερη. Γιατί? Ενώ είχαμε τη διαπραγματευτική ομάδα ε, δίπλα στην Κομισιόν και κάναμε διαπραγματεύσεις και παίρναμε ας πούμε ειδήσει ας πούμε σε πραγματικό χρόνο για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων για να θέσει συναντήσει με τον Υπουργό. Ε, Εποφεληθήκαμε λοιπόν από την παρουσία του, του Υπουργού, για να κοιτάξουμε και τις εμπορικέ σχέσεις και την ε, εμπορική πολιτική του Μεξικού που είναι πάρα πολύ δραστήρια και ενεργή και να εξετάσουμε το συνεγγύ στι πρόσφατε μεταρρυθμίσει στο Μεξικό σε βασικού τομεί τη οικονομία, που δημιουργούν και πολλέ ευκαιρίε και για ευρωπαϊκέ εταιρείε. ε, δεδομένης δυνατότητας αναβάθμισης της ε, συμφωνίας. Τώρα, το Μεξικό είναι τμήμα των διαπραγματεύσεων του TTIP. Ε, ε, διαπραγματεύονται με την Τουρκία, η Ορδανία, έχουν συνάψει πρόσφατα ε, συμφωνία με την ε, Χιλή, Οικονομική, ε, Κολομβία και Περού. Δεν θέλουν να χάσουν αυτές τις σημαντικές διαπραγματεύσεις με εμά. Ε, είμαστε σημαντικός κρίκος. Ο Υπουργός είπε ότι θέλει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις μαζί μας για τον εξυγχρονισμό της εμπορικής συμφωνίας και λόγω του TTIP βέβαια. Ε, θα υπάρχει μια δυνατότητα, ας πούμε, μια άλλη οδός, μια άλλη ατραπός, ας πούμε, αν ολοκληρωθεί το TTIP. Και θα υπάρχει και η ΣΥΤΑ που θα επικυρωθεί σύντομα. Επομένως, έχει μια ευκαιρία το Μεξικό να αναβαθμίσει την συμφωνία με εμά. Και το είπε μάλιστα ειλικρινά, γιατί είναι αυτό ασύνηθες. Συνήθω οι, οι αξιωματούχοι του Μεξικού δεν μιλάνε τόσο ανοιχτά και ειλικρινά. Ε, διατρέξαμε τις βασικές μεταρρυθμίσεις που έκανε το Μεξικό στην ενέργεια, στο τομέα της ενέργειας. Ε, μια, έχουμε μια τεράστια προγράμματα δημοσίων προμηθειών στο Μεξικό. Είναι έτσι, στο pipeline. Έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν οι δικές μας εταιρείες, οι ευρωπαϊκές, να είναι πιο δραστήριες στον τομέα αυτό στο Μεξικό. Και επίσης εξετάσαμε τον, τη μεταρρύθμιση του, τομέα των τηλεπικοινωνιών, που για πρώτη φορά ε, σταμάτησε το ιστορικό μονοπόλιο που είχε στο Μεξικό η κρατική εταιρεία και έχουν δυνατότητα και οι ξένες εταιρείε ε, να παίξουν σε αυτή την αγορά, κυρίως οι Αμερικάνικες το κάνουν ήδη. Ήταν ε, μια πολύ ενημερωτική και ειλικρινής ε, ανταλλαγή απόψεων. Η επίσκεψη του Υπουργού ήταν κρίσιμη στα πλαίσια της διαδικασίας ολοκλήρωσης της αποτίμης κατάστασης, το scoping exercise. Και στις 12 Ιουνίου, ε, την τελευταία μέρα της ε, Συνόδου Κορυφής με το Μεξικό, είχε αναγγελθεί η έκθεση ε, ήταν Μιλούσα για τα βασικά εμπόδια που υπήρχαν στην ολοκλήρωση της συμφωνίας και τώρα η Κομισιόν τελειώνει την μελέτη αντικτύπου και θα, σύντομα θα ζητήσει ε, τη διαπραγματευτική εντολή. Οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν στα τέλη του 2015 ή στις αρχές του 2016. Σχόλια όχι. Άρα, υπάρχει πρόοδος. υπάρχει δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα νέο μέτωπο, ένα νέο μέτωπο σχέσεων. Η Ιαπωνία. Ε, με επαφές είχαμε στις 12 Μαΐου. Ο κ. Πετριτσόνε ήταν ο βασικός διαπραγματευτής. Έχω την ενημέρωση ότι και στο μέτωπο της ε, Ιαπωνίας υπάρχει πρόοδος και κατά πάσα πιθανότητα η ολοκλήρωση τη εμπορική Συμφωνία ευρωπαϊκή Ένωση ή ε, Ιαπωνίας να λάβει χώρα στο τέλος του 2015. Ε, Καναδάς. Συνάντηση 3 Μαρτίου και 5 Μαΐου. Με βασικό πραγματευτή τον κύριο Φορσίτερ και τον πρέσβη του Καναδά στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρόντα και τον κύριο Πετριτσόνε που ήταν επίση ε, βασικό διαπραγματευτή και στην περίπτωση του Καναδά. Δουλεύει πολύ αυτό ο κύριο. Στι 15 Ιουνίου, χθε δηλαδή, έγινε μια άλλη συνάντηση με τους Καναδούς. Ο κύριος Πάπριξ δεν είναι εδώ. Ήσασταν παρόν. Άρα δεν έχουμε άλλες προφορίες για το θέμα του Καναδά. Ήταν κάποιο από εσά παρόν ε, στη συνάντηση με τι Καναδικέ αρχέ. Όχι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί, γιατί αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα θα το είχαμε ακούσει. Και περνάμε στο σημείο 19 της Μέσης διάταξη. διάταξης, έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με θέμα τα εμπόδια στο εμπόριο και τις επενδύσεις, έκθεση του 2015. Δίνω το λόγο στον κύριο Σορμέλης. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την πέμπτη εκδοχή Τη έκθεση για του εμπορικού και επενδυτικού φραγμούς που υιοθετήθηκε από την Κομισιόν στις 17 Μαρτίου και παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου. Όπως και τα προηγούμενα έτη, η έκθεση κάνει μια επισκόπηση καταρχάς των ε, συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων ε, για τέτοια θέματα, ε, κατά απαριθμεί τα βασικά εμπόδια που έχουν οι έξι στρατηγικοί οικονομικοί εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η Κίνα, η Ινδία, η Ιαπωνία, Μέρκοσουρ, όπου εξετάμε, εξετάζουμε κυρίως τη Βραζιλία και την Αργεντινή Ρωσία και οι Ηνωμένε Πολιτείες. Από την αρχή αυτής της έκθεσης αυτός ήταν, ε, αυτό ήταν το γεωγραφικό εύρος το οποίο καλύπτουμε. Και η έκθεση επίσης έχει και ένα τρίτο τμήμα που μιλάει για τις διαφορετικές στρατηγικές που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει τους βασικούς φραγμούς. Ο στόχος της έκθεσης είναι να υπάρξει αφύπνιση και συνειδητοποίηση σε πολιτικό επίπεδο ε, για τα πιο σημαντικά εμπορικά προβλήματα και φραγμούς και να μιλήσει για τη σημασία του να αντιμετωπιστούν συντονισμένα αυτά τα εμπόδια και τροχοπέδες. Γι' αυτό στην έκθεση εστιάζουμε στις βασικές προτεραιότητες μόνο, δηλαδή τις προτεραιότητες που αφορούν την πρόσβαση στην αγορά. Και η έκθεση είναι συμπληρωματική προς μια ευρύτερη έκθεση που ετοιμάζουμε, την έκθεση παρακολούθησης του προστατευτισμού, που ετοιμάζουμε τη ΣΥΟΣ και που αποτελεί ένα πιο λεπτομερές κείμενο ε, για τα, τους φραγμούς που έχουν διάφορες χώρες. Επομένως αυτές οι δύο εκθέσεις είναι συμπληρωματικές. Οι διάφορες περιπτώσεις που συμπεριλάβαμε σε αυτή την εκδοχή της έκθεσης είναι 28. Η Ρωσία είναι πάνω-πάνω με 7 περιπτώσεις ε, φραγμών ε, πρόσβαση στην ε, αγορά, η Κίνα έξι περιπτώσεις και τέσσερι ε, υποθέσεις έχουμε για την Ινδία και την Βραζιλία, τρεις υποθέσεις για την Αργεντινή και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ιαπωνία είναι ειδική περίπτωση, γιατί ξανά περιγράψαμε τους φραγμού στην έκθεση στα πλαίσια της ε, συνεχιζόμενης διαπραγμάτευσης για την Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου, ε, που δικαιολογούνται από το συγκεκριμένο πλαίσιο για τις μη δασμολογικές ποσοστώσεις. Τον κατάλογο με, το, με τους φραγμούς αυτούς το στείλαμε στην Ιαπωνία στα τέλη του 2014. Ε, συχνά οι φραγμοί αυτοί αφορούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ε, τα θέματα φυτογενομικής προστασίας, ε, και τοπικού περιεχομένου. Απαιτήσει τοπικού περιεχομένου. Για ε, αυτό το τρίτο. Έχουμε διακριτική φορολόγηση σε διάφορους τομείς στην Βραζιλία ας πούμε. Άλλα σημαντικά παραδείγματα είναι το νέο, ο νέος νόμος ε, της Ρωσίας για την, τον εντοπισμό προσωπικών δεδομένων που απαιτούν όλα τα δεδομένα ε, Ρώσων πολιτών να αποθηκεύονται και να τυχάνουν επεξεργασία στη Ρωσία. Αυτό ε, θέλουν να το υιοθετήσουν ε, και άλλες τρίτες χώρες για το τοπικό περιεχόμενο. Ε, επίσης, διάφορα μέτρα έχουν επιβάλει οι κινέζικες αρχές στο τομέα της ε, ασφάλεια. Αυτό δεν το απεικονίζουμε καλά στην έκθεση γιατί είναι καινούριο. Ε, φυτογενομικά εμπόδια στην Βραζιλία έχουμε, στην Κίνα, στι Ηνωμένες Πολιτείες και στη Ρωσία. Και θέματα IPR ε, αναφέρονται στην έκθεση και αφορούν την Κίνα και τι Ηνωμένε Πολιτείε, Το UGIs, θέμα που συζητάμε στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για το TTIP. Επίσης, μιλάμε για θέματα επενδύσεων και θέματα ιδιοκτησία στην Βραζιλία, ε, για τους περιορισμούς της Κίνας στις ξένες επενδύσεις, που δημιουργούν ε, ανησυχίες, παρά το γεγονός ότι έχει κάνει κάποιες μεταρρυθμίσεις η Κίνα, κυρίως ε, την πιλωτική την ε, ζώνη ελευθέρου εμπορίου που έχει δημιουργηθεί γύρω από τη Σανγκάη και που το, το δοκιμάζουν οι Κινέζοι πιλωτικά. Για πώς αντιμετωπίζουμε τα, τους φραγμούς αυτούς. Χρησιμοποιούμε τις διαπραγματεύσεις ε, για συμφωνίες ε, ελευθέρου εμπορίου. Έχουμε τέτοιες διαπραγματεύσεις με τέσσερις από τους έξι στρατηγικούς εταίρους. Ε, καθώς και διαπραγματεύσεις για τα επενδυτικά θέματα αυτή τη στιγμή που κάνουμε με την Κίνα. Επίσης, ε, εφαρμογή και παρακολούθηση των ε, συμφωνιών που υπάρχουν μέσω της στρατηγικής πρόσβασης στην ευρωπαϊκή αγορά. Τρίτον, χρησιμοποιούμε το, τη διαδικασία επίλυση των διαφορών του ΠΟΕ όταν είναι κατάλληλο αυτό και σε διάφορες περιπτώσεις περνάμε μέσω του ΠΟΕ. Ας πούμε, όπως στη Ρωσία. Τρει από τις 7 υποθέσεις που είχαμε με τη Ρωσία ανοιχτέ πέρασαν από εκεί. Μέσω του ΠΟΕ, δηλαδή του Μηχανισμού επίλυση Διαφορών. Τέταρτος τρόπος που έχουμε είναι οι επιτροπέ του ΠΟΕ. Εμείς είμαστε από τα πιο ενεργά μέλη, κυρίως στην TPT και στο SPS και στην Επιτροπή TRIMS. Τέλος, έχουμε και διμερείς και πολυμερείς διεθνείς συνόδους κορυφής, όπου εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση οι μεμονωμένα κράτη-μέλη συμμετέχουν. Για να ολοκληρώσω λοιπόν αυτή την έκθεση, από την έκθεση φαίνεται ότι οι στρατηγικοί μας εταίροι έχουν μία πλειάδα ε, φραγμών που είναι δύσκολο να τα αντιμετωπίσουμε, πολλών και διαφορετικών. Σίγουρα χρειαζόμαστε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα σε πολιτικό επίπεδο και πιο καλή εφαρμογή της στρατηγικής πρόσβασης ε, των τρίτων χωρών ε, στην ευρωπαϊκή αγορά για να μπορέσουμε να καταρρύψουμε τους φραγμούς. Αυτές οι προσπάθειες δεν μπορούν να γίνουν μόνο από την Κομισιόν, σίγουρα. Θα πρέπει να εμπλέκουν και τα κράτη-μέλη μέσω των συναντήσεων υψηλού επίπεδου και μέσω του δικτύου πρεσβειών που έχουν στις εν Αυτές οι προσπάθειες επίσης θα πρέπει να εμπλέκουν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν ε, οι ευρωβουλευτές έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν αυτές τις τρίτες χώρες και όταν μπορούν να διαμηνήσουν πολιτικά μηνύματα σε υψηλό επίπεδο στις αρχές των χωρών αυτών. Φυσικά είμαστε έτοιμοι να σας δώσουμε τα στοιχεία, τα απαραίτητα στοιχεία και τα μηνύματα κατάλληλα, ούτω ώστε να μιλήσετε για αυτού τους εμπορικούς φραγμούς, ε, τους οποίους αναφέρει η έκθεση. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ, δεν μου έχει ζητήσει και το λόγο. Α, ο Χέλμουτ. Μπορούμε να έχουμε την έκθεση σε γραπτή μορφή. Γιατί τα νούμερα που αναφέρατε και οι περιπτώσεις παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Θέλουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό, αλλά αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε να έχουμε το έντυπο σε γραπτή μορφή την έκθεση αυτή. Ο Πρόεδρος νομίζω ότι έχει κυκλοφορήσει, αλλά θα σας τη διανύμουμε και πάλι. Επιτρέψτε μου τρία ερωτήματα να διατυπώσω. Πρώτον, Στην τελευταία δημόσια μορφή του, η φόρμα του ΠΟΕ, μάλλον στην τελευταία δημόσια ενημέρωση του ΠΟΕ, υπήρξε δήλωση και ενημέρωση για τα εμπόδια στο εμπόριο και κατά πόσο έχουν αυξηθεί ή μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Αναφέρεται μια χώρα εκεί και την αναφέρατε κι εσείς. Και εσείς το πιστεύετε αυτό, ότι δηλαδή τα μέτρα που είναι κατά του εμπορίου και των επενδυτικών ροών έχουν αυξηθεί. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες που εξηγούν αυτή την αύξηση. Αυτό καταρχάς. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση πλήττεται από αυτή την αύξηση κατά μέσο όρο. Η, η αύξηση αυτών των μέτρων στρέφεται συγκεκριμένα εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τρίτον, υπάρχει διαφορά στα εμπόδια τα εμπορικά σε σχέση με τα προϊόντα εξαγωγών και την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού. Δηλαδή τα εμπόδια βεβαίως πλήττουν τα προϊόντα που εξάγονται σε ένα πρώτο επίπεδο, αλλά σε ένα δεύτερο επίπεδο ακόμα μεγαλύτερο πλήγμα θα υποστεί η παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, προσφοράς αν θέλετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για το πρώτο σας ερώτημα να πω ότι πράγματι στην ανάλυση που κάνουμε διαπιστώνουμε ότι συνολικά αυξάνονται τα εμπορικά εμπόδια, οι φραγμοί σε αυτό δεν, είναι ένα θέμα που δεν αναπτύσσουμε περιστατωμένα στην έκθεση γιατί έχουμε επιλεκτικά διαλέξει κάποιες περιπτώσεις μόνο. Ωστόσο, το ύψος του προστατευτισμού δείχνει ότι κάθε χρόνος που περνάει ε, σηματοδοτεί και προσθήκη τέτοιου είδους μέτρων, ε, ό,τι προστίθεται δεν αντισταθμίζει ε, ε, διαγραφή παλαιότερων ή εξάλληψη παλαιότερων, γιατί αυτό το δεύτερο σκέλος δεν γίνεται. Άρα, αθρηστικά έχουμε αύξηση, ναι. Και αυτό είναι λόγος ανησυχίας. Από εκεί και πέρα. Έχουμε ξεκινήσει αυτή την άσκηση παρακολούθησης στο πλαίσιο της μακροοικονομικής κρίσης και βλέπαμε ότι σε περιοχές που έβγαιναν από κρίση μειωνόταν αυτή η τάση. Όμως, όσες χώρες έχουν ε, ε, επιβάλει τέτοιου είδους εμπόδια και φραγμούς, ε, τότε στον καταστατικό τους χάρτη, να το πω έτσι, η τάση αυτή δεν είναι μειωτική. Έχουν την τάση τα μέτρα αυτά να παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και πέρα και μετά την κρίση αν θέλετε. Τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λέω ότι τα μέτρα στοχεύουν συγκεκριμένα και απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν γίνει επισκοπού επί τούτου. Όμως αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο βασικός εταίρος πολλών εταίρων, πολλών άλλων χωρών και πιο συγκεκριμένα του γείτονα εξ Ανατολών, τότε ναι, τέτοιου είδου περιοριστικά μέτρα και φραγμοί έχουν αντίκτυπο περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά σε άλλου εταίρου που συναλλάσσονται με τη συγκεκριμένη χώρα. Τρίτον, οι περιορισμοί στις εξαγωγές. Είδαμε επανειλημμένος αύξηση της έγκρισης των περιορισμών στις εξαγωγές. Και αυτό είναι ανησυχητικό φυσικά. γιατί δείχνει ένα είδος εθνικισμού ως προς τους πόρους. Κάποιες χώρες θέλουν να διατηρήσουν τις πρώτες ύλες, ύλες προς όφελος της εχώριας βιομηχανίας ε, ε, με, της μεταποιητικής. Και αυτό είναι κάτι που εμείς καταπολεμούμε. Στη διμερή ατζέντα προσπαθούμε να εξαλειφθούν ε, οι περιορισμοί στις εξαγωγές και οι εξαγωγικοί δασμοί ε, σε όλες αυτές τις συμφωνίες που έχουμε με τρίτες χώρες. Είναι δύσκολο να πετύχουμε τέτοια αποτελέσματα γιατί το βιβλίο με τους κανόνες στην πολυμερή ε, ε, συμφωνία είναι πιο αδύναμο από τους περιορισμούς της εξαγωγές που εφαρμόζουν οι πιο οι τρίτες χώρες. Αλλά, μπορούμε, αλλά προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο φιλόδοξοι. και είναι αυτό προτεραιότητα για εμάς, όχι μόνο στις διμερείς διαπραγματεύσεις, αλλά και ε, στο πλαίσιο ε, των διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση στον ΠΟΕ, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Και βέβαια ε, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την πρόσβαση στην αγορά. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση. Μας διευκολύνει ιδιαίτερος στη δουλειά μας στην Επιτροπή θα παραμείνουμε σε επαφή για το υπόλοιπο της χρονιάς ασφαλώς. Και τον επόμενο γύρο, το επόμενο επεισόδιο θα έρθετε να μας το παρουσιάσετε στην ε, Επιτροπή μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχει αναβληθεί η συζήτηση για το σημείο 20 και το σημείο 6 που θα αντικαθιστούσε το 20 αναβλήθηκε η συζήτηση και γι' αυτό. Θα έχουμε λοιπόν στις 29 Ιουνίου συζήτηση στην Επιτροπή μας για την Ενεργειακή Ένωση. Έρχομαι λοιπόν στο σημείο 21. Υπό τα διάφορα. Υπάρχει κάτι που θέλετε να θέσετε υπό τα διάφορα. Βλέπω πως όχι. Άρα, επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας θα λάβει χώρα στις 29 Ιουνίου της φετινής χρονιάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.